Um, we're just going to... Um, Καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρία. Παρακαλώ, καθίστε. Αυτή είναι η τελευταία μας συνάντηση για αυτό το διήμερο. καλωσορίσατε. Όπως γνωρίζατε, είχαμε μια εξέντηση από τα μέλη σήμερα. Και κάποιοι νομίζω ανησυχούν για το καιρό, αλλά παρόλα αυτά έχουμε κάποιους σημαντικούς συναδέλφους εδώ, οι οποίοι καλό είναι που βρίσκονται εδώ και είμαι σίγουρο θα κάνουν δύσκολες ε, ερωτήσεις ε, και τους καλωσορίζω στη συνάντησή μας, καλωσορίζω επίσης και όσους μας ε, παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Όπως θα γνωρίζετε, ο κ. Καλέχα είναι τώρα Γενικός Διευθυντής της ε, Γενικής Διευθύνσης Επιχειρήσεων. Δεν είναι ξένος στο Κοινοβούλιο, διότι τον έχετε συναντήσει πολλοί από εσάς όταν ε, δούλευε στο γραφείο της κυρίας Δεπλάσιο, καθώς και στη, ε, υπήρξε και υπάλληλος Κομισιόν για πολύ καιρό. Είναι κάποιο που εκτιμά ιδιαίτερα την πολιτική διαδικασία και ήθελε να έρθει να μα μιλήσει εδώ και καιρό και επιτέλου καταφέραμε. Θα μα μιλήσει για το μελλοντικό πρόγραμμα εργασία τη γενική διεύθυνση Επιχειρήσεων. Ουσιαστικά το έργο που θα έχουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος πιθανώς της θητείας αυτής ε, του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν διότι βρισκόμαστε στους τελευταίους 18 μήνες. Επίσης, ε, του ζήτησα να μας μιλήσει για τις εξέλιξει τη ε, Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι γνωρίζω ότι εμπλέκεται ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων στον κανονιστικό διάλογο και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την παρούσα Επιτροπή, όπω γνωρίζετε. Και πολλοί από εμάς ταξίδεψαν στη Washington πέρυσι και ήμασταν σε επαφή με του Αμερικανου. Ε, την ρυθμιστική μονάδα της Αμερικής για διεθνή συνεργασία σε οδομέτρα ηλεκτρικών, των ηλεκτρονικών και έχουμε οργανώσει κάποιε διασκέψεις για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα να συζητήσουμε. Σας δίνω λοιπόν κύριε Καλέχα το λόγο και μετά θα λάβουν το λόγο τα μέλη για να σας κάνουν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάλκομ Χάουρμπορ, αξιότιμα μέλη, με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ μπροστά στην Επιτροπή σας. Ήθελα να... Είχα έρθει πριν τα τέλη του 2012, αλλά χαίρομαι που τελικά τα καταφέρνω πριν από το τέλη Ιανουαρίου του 2013. Διότι, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Πρόεδρος, η φετινή χρονιά θα είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο λόγος είναι ότι εισερχόμαστε στην τελική περίοδο αυτής της θητείας και αυτής της Επιτροπής. Και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Αυτή η δουλειά θα λάβει χώρα σε μια πολύ σημαντική και δύσκολη εποχή της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω την οικονομική κρίση και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει στις βιομηχανίες μας. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση στην Ευρώπη, χάσαμε 3 εκατομμύρια θέσει εργασία στη βιομηχανία. Η βιομηχανική μας παραγωγή έχει μειωθεί κατά 10%. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι πολύ χαμηλή. Και επίσης παρατηρήσαμε μείωση της μεταποίησης και της ανταγωνιστικότητας. Ως Γενικός Διευθυντής λοιπόν των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας και υπογραμμίζω το και της βιομηχανίας έχουμε μια σημαντική προτεραιότητα μπροστά μας. Η προτεραιότητα κλειδί είναι να ανακτήσουμε ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Έδειχνα στον κύριο Μάλκολμ Χάρμπορ το λογότυπο τη φιλοδοξία της ε, γενικής μας διεύθυνσης που είναι ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και το ερώτημα είναι πώς θα το επιτύχουμε. Ο μόνος τρόπος είναι να θέσουμε την πραγματική οικονομία στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Για πολλά χρόνια λέγαμε ότι η καλύτερη βιομηχανική πολιτική είναι η ανύπαρκτη βιομηχανική πολιτική ή ότι η βιομηχανική πολιτική αφορά το να επιλέγει κανείς ε, τους νικητές και τους ιτημένους και να επιχορηγεί. Εμείς θεωρούμε ότι και οι δύο αυτές προσεγγίσεις είναι λανθασμένες. Χρειάζεται να αναπτύξουμε στην Ευρώπη μια νέα στρατηγική βασισμένη στην πραγματική οικονομία και στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας των διαφόρων τομέων. Να βασίζεται επίσης ε, σε μια δυναμική πολιτική για τις μικρόμεσες επιχειρήσεις, διότι αυτό είναι ουσιώδους σημασία. Επίσης πρέπει να εστιαστούμε σε μέσα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο αυτήν την ανανεωμένη στρατηγική που ονομάζουμε επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Reindustrializing Europe, ο κ. Σταγιάννη, σε την παρουσίασε τον Νοέμβριο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να σας ενημερώσω ότι οι Υπουργοί στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας επικύρωσαν τη στρατηγική το Δεκέμβριο και επικύρωσαν τον στόχο που εμείς έχουμε θέσει. Ο στόχος αυτός είναι να είμαστε βέβαιοι ότι το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕΠ θα ανέρχεται σχεδόν στο 20% έως το 2020. Προσθέσαμε και ένα τέταρτο εικοσαέρι σε αυτή τη στρατηγική 2020. Δεν θα είναι μόνο 20% λιγότερες εκπομπές ρήπων, δεν θα είναι μόνο 20% περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 20% μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να φροντίσουμε η βιομηχανία να φτάσει στο 20% του ΑΕΠ. Είναι δυνατό. Αυτή τη στιγμή η βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 15,5% του ΑΕΠ. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα πρέπει να καταβάλουμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια, διότι μέσω της βιομηχανίας του τομέα της μεταποίησης θα παρέχουμε και υπηρεσίες, θα συνδυάσουμε την παραγωγή με τις υπηρεσίες για να μπορέσουμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Αυτή η χρονιά, το 2013, ξεκίνησε με άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία στις 9 Ιανουαρίου. Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα. Για να βγούμε από την κρίση, χρειαζόμαστε επίσης περισσότερους επιχειρηματίες στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή σημειώνεται μεγάλη μείωση της επιχειρηματικότητας στην Ήπειρό μας. Στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ασία αντιθέτως πάνω από τους μισούς νέους που έχουν ερωτηθεί λένε θέλω να είμαι ελεύθερος επαγγελματία, θέλω να φτιάξω τη δική μου επιχείρηση. Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 37% μόλις και πριν από τρία χρόνια ήταν 45%. Εάν δεν παρέμβουμε θα χάσουμε μια ολόκληρη γενιά επιχειρηματιών. και θα έχουμε δημιουργήσει μια τεράστια στρατηγική. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια στρατηγική που να καλύπτει όλους τους τομείς. Αυτό που θα ήθελα να σας ε, πω σήμερα είναι ποιες θα είναι οι κύριες προτεραιότητες για το 2013 στο πρόγραμμά μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι οι τρεις πρωτοβουλίες θα πρέπει να θεωρηθούν στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος και θα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της Επιτροπής σας, διότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με 500 εκατομμύρια καταναλωτές στην εξάλληψη των τελευταίων φραγμών για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών παραμένει σημείο κλειδί της στρατηγικής μας. Θα ήθελα λοιπόν να, να οργανώσω την παρουσιασή μου με βάση τρία κύρια μέρη. Τα τρία στοιχεία αυτά που θα ήθελα να αναπτύξω είναι πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι οριζόντιες στρατηγικές που αφορούν την νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς και που θα, θα συζητήσουμε και θα προτείνουμε. Δεύτερον, τυποποίηση. Τρίτον, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες τομέακες πρωτοβουλίες. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις οριζόντιες πρωτοβουλίες για την νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς. Εδώ έχουμε ένα εργαλείο κλειδί, το οποίο μερικές φορές λησμονούμε. Είναι η οδηγία 9834. Αυτή η οδηγία επιβάλλει στα κρατημέλη να κοινοποιούν στην Κομισιόν και στα λοιπα κράτη-μέλη όλους τους εθνικούς ε, τεχνικούς κανονισμούς, τα σχέδια τεχνικών εθνικών κανονισμών για προϊόντα και για τις υπηρεσίες της κοινωνικής πληροφοριών πριν υιοθετηθούν στην εθνική νομοθεσία. Έτσι μπορούμε να παρέμβουμε ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία φραγμών. Το 2012 η Κομισιόν εξέδωσε 64 λεπτομερείς γνωμοδοτήσεις, 150 σχόλια. Σταματήσαμε μια σειρά πρωτοβουλειών διότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να αποφύγουμε νέους φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Σε θέματα νομοθεσίας, για τα εναρμονισμένα και τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, η εσωτερική αγορά για τα αγαθά υπάρχει. Έχει καθιερωθεί, αλλά χρειάζεται περισσότερη επιβολή. Η επιβολή είναι κάτι σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε σωστά το κοινό συμφέρον και να διασφαλίσουμε ότι το εμπόριο θα πραγματοποιείται από δίκαιε και σωστέ επιχειρήσει σε ασφαλή συνθήκε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά επίση και την προστασία των καταναλωτών. Μόνο ασφαλή προϊόντα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά. Διαφορετικά, οι καταναλωτέ μα θα απολέσουν εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά. Γι' αυτό τον λόγο, μέσα στι επόμενε ημέρε, η Κομισιόν θα εγκρίνει ένα νέο πακέτο ασφάλειας προϊόντων στην αγορά και επιτήρησης της αγοράς και της ασφάλειας. Το τονίζω διότι θα αναθεωρήσουμε τη γενική, το γενικό κανονισμό ασφάλειας των προϊόντων και θα έχουμε ένα νέο μέσο επιτήρησης της αγοράς με πολιετές σχέδιο δράσης για την επιτήρηση της αγοράς. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού, στις δέσμες μέτρων αυτού του πακέτου, σκοπός είναι να υπάρξουν σαφείς απτές βελτιώσεις στην δυνατότητα επιβολής της ε, νομοθεσίας της Ένωσης για τα προϊόντα. Αυτό αποτελεί κομμάτι τόσο της πραξενίας αγοράς και της βιομηχανικής πολιτικής. Πρέπει να επιβάλλουμε το σύστημα επιτήρησης των αγορών ώστε να αποφύγουμε την ύπαρξη μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων αγαθών στην αγορά. Πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργία του παρόντο συστήματο επιτήρηση των αγορών στην Ευρώπη. Αυτό θα το κάνουμε δημιουργώντα ένα πλαίσιο επιτήρηση των αγορών ενό επίπεδου που αναφέρεται σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ένα ψήφισμα που προετοίμασε η δική σα επιτροπή. Εκεί εμεί θα εισάγουμε διάφορε απλουστεύσει, θα ξεφορτωθούμε διάφορε επικαλύψει, θα μειώσουμε τι ανάγκε κατηγοριοποίηση των προϊόντων στο ελάχιστο και θα προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τους κανόνες για όλα τα προϊόντα στο βαθμό του δυνατού. Έτσι θα είναι πιο ομοιόμορφη η εφαρμογή της επιβολής ε, της επιτήρησης των αγορών σε όλα τα κρατημέλη. Θα υπάρχει καλύτερη προστασία για τους καταναλωτές, πιο ομοιόμορφες συνθήκες εμπορικών συναλλαγών για τους οικονομικούς φόρους και λιγότερος οικονομικός φόρτος. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα την λάβετε μέσα στο μήνα Φεβρουάριο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξέρουμε ότι δεν μένει πολλής χρόνο θητείας, αλλά ελπίζουμε ότι η παρούσα Επιτροπή θα αφιερώσει χρόνο σε αυτό το μέσο ω σημαντική προτεραιότητα γιατί θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για την ενίσχυση τη εσωτερική αγορά. Η δεύτερη πρωτοβουλία που εξετάζουμε είναι η επιθεώρηση τη εσωτερική αγορά για τα βιομηχανικά προϊόντα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απλωστεύσουμε και να εξυγχρονίσουμε τους σημερινούς κανόνες της ενιαίας αγοράς. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Ελέγχουμε κατά πόσο η νομοθεσία μας είναι ενημερωμένη, επικαιροποιημένη, βάσει των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων. Ορισμένοι από τους κανόνες αυτούς είναι πλέον πεπαλαιωμένοι και χρειάζεται να τους επικαιροποιήσουμε βάσει των σημερινών στοιχείων τη σημερινή πραγματικότητα. Ο δεύτερο στόχο που επιδιώκουμε είναι η νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη την παγκοσμιοποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τι τελευταίε κατασκευαστικέ πρακτικέ και εξελίξει στην αλυσίδα παραγωγή και προμηθειών. Η τρίτη προσέγγιση, αν υπάρχουν ακόμα φραγμοί στο εσωτερική αγορά που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσουμε ώστε η νομοθεσία να είναι στο ύψος των νέων εξελίξεων. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική δέσμη μέτρων, πριν δύο μέρες ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση προς όλους τους οικονομικούς τομείς και ρωτάμε από οργανισμούς φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, πείτε μας ποιοι είναι οι φραγμοί που έχετε εσείς αντιμετωπίσει στις καθημερινές σας συναλλαγές. Πείτε μας, σε ποια σημεία δεν έχει επικαιροποιηθεί η νομοθεσία. Πείτε μας, ποια είναι τα θέματα που εσείς θεωρείτε ότι χρειάζονται διόρθωση. Και χρησιμοποιούμε αυτή τη διαβούλευση επίσης για να κάνουμε και μερικές ερωτήσεις. Όσον αφορά νέους τομείς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τις, τι, ε, e, τις ε, βασικές τεχνολογίες και enabling technology εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με κάποιο τρόπο, με τεχνογνωσία. Θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτή τη διαβούλευση μέσα στου επόμενου μήνε και βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, σκοπό είναι να παρουσιάσουμε μια πρωτοβουλία απλούστευση τη εσωτερική αγορά για τα βιομηχανικά προϊόντα, εξαλείφοντα φραγμού και εμπόδια. Επίση, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι σε σχέση με Μαζί με αυτή την πρωτοβουλία θα κάνουμε έναν έλεγχο καταλληλότητας της υπάρχουσας νομοθεσίας από τον οποίο έλεγχο θα λάβουμε στοιχεία για να βελτιώσουμε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερη λοιπόν πρωτοβουλία μαζί με την επιτήρηση των αγορών, απλούστευση της εσωτερικής αγοράς για τα βιομηχανικά προϊόντα. Τρίτος τομέας εργασίας, ορισμένες συγκεκριμένες οδηγίες. Πρέπει να συνεχίσουμε με τι οδηγίε που αφορούν συγκεκριμένου τομεί και το 2013 και ξέρω ότι η παρούσα επιτροπή ακολουθεί ενδελεχώς τα διάφορα στοιχεία. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα κείμενα για τον ατομικό προστατευτικό ε, εξοπλισμό, ε, σωσίβια, ε, κράνη, εξοπλισμό για φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Γιατί παρουσιάζουμε αυτά τα κείμενα εντάσσονται στη διαδικασία εναρμόνισης της νομοθεσίας στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Μοιάζει η προσέγγιση με τη δεσμή μέτρων ευθυγράμμισης που εσείς διαπραγματεύεστε αυτή τη στιγμή με το Συμβούλιο. Αποτελεί σημαντικό βήμα προς την απλοποίηση των κανόνων της εσωτερικής αγοράς και την ελάττωση των διοικητικών φόρτων για την ασφάλεια. Σκοπός είναι να ενισχυθεί το σύστημα από άποψη ασφάλειας προϊόντων και η βελτίωση της επιτηρήσης των αγορών καθώς και ταυτόχρονα ελάττωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις μας. Και καθώς μιλάμε για μείωση του διοικητικού φόρτου, θα ήθελα να κλείσω αυτό το πρώτο κεφάλαιο με ένα τέταρτο στοιχείο. Ίσως δεν έχετε αντιληφθεί ότι μάθει ότι ξεκινήσαμε πριν τα Χριστούγεννα και άλλη μία δημόσια διαβούλευση για τις δέκα πιο επαχθείς νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πείτε μας ποια νομοθετικά κείμενα είναι πλέον επαχθή για εσάς. Έλαβε η Κομισιόν πάνω από χίλιες απαντήσεις από επιμέρους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από επαγγελματικούς οργανισμούς, η γενική μας διεύθυνση ήταν ο τυχερός νικητής. Τώρα ε, ταξινομούμε για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τα 10 χειρότερα νομοθετικά κείμενα που υπάρχουν. Θα τα δημοσιεύσουμε. Θέλουμε να τα συζητήσουμε. Θέλουμε να τα παρουσιάσουμε. Δεν το κάνουμε απλά για να φτιάξουμε μια ταξινόμηση, έναν κατάλογο. Φυσικά βάσει των όσων διαπιστωθούν θα αναζητήσουμε βελτιώσεις για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Μπορώ ήδη να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτά τα νομοθετικά κείμενα περιλαμβάνονται και νομοθεσίε τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Θα ζητήσω λοιπόν στου συναδέλφου να δουλέψουμε σκληρά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε βελτιώσει. Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι εξαιρετικά σημαντική. Πρέπει να δείξουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίε μα. Και πρέπει εγώ να σα πω ε, ω εντεταλμένο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και ω γενικό διευθυντή, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτό το τομέα. Σε αυτές τις εποχές δύσκολης λιτότητας πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μειώσουμε το κόστος επιχειρηματικών συναλλαγών, απλούστευση και η μείωση της γραφειοκρατίας είναι εξαιρετικά σημαντική γι' αυτό. Θα σας πω και μερικά καλά νέα. Ζητήσαμε επίσης να μάθουμε από τις επιχειρήσεις. Τους ρωτήσαμε, μπορείτε να μας πείτε ποια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλή. Και η πρώτη απάντηση που λάβαμε η καλύτερη απάντηση ήταν η οδηγία για τις καθυστερημένων πληρωμών που προέρχεται από εσάς και θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την παρούσα Επιτροπή διότι ε, χάρη στην εξαιρετική δουλειά των δικών σας μελών καταφέραμε να επιτύχουμε αυτή την οδηγία. Ωστόσο, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Απομένει κάτι ακόμα πολύ σημαντικό να κάνουμε φέτος όσον αφορά αυτή την οδηγία καθυστερημένων πληρωμών. Αλλά είναι πραγματικά, ε, σύμφωνα με τις απαντήσεις, η καλύτερη νομοθεσία που έχουμε φτιάξει. Ε, ας μιλήσουμε τώρα για την τυποποίηση και τις διάφορες ε, ε πρωτοβουλίες. Πέρυσι το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο ενέκρινε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Τυποποίησης. Αποτελεί ορόσημο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τα πρότυπά της. Τα πρότυπα μειώνουν το κόστος για τις επιχειρήσεις, αλλά αποτελούν και κρίσιμο παράγοντα που ενισχύει τον ανταγωνισμό. Εμείς, ενισχύοντας το σύστημα τυποποίησής μας, μπορούμε να καταλήξουμε και σε παγκόσμια πρότυπα. Θα μπορούσαμε να είμαστε ηγέτες σε αυτό το τομέα και αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ο νέος κανονισμός τώρα χρειάζεται να υλοποιηθεί και φέτος εμείς θα παρουσιάσουμε μέσα στους επόμενους μήνες, γίνονται αυτή τη στιγμή εργασίες, για πρώτη φορά θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τυποποίηση ένα νέο εργαλείο επικοινωνίας για την αύξηση της διαφάνειας των μελλοντικών εντολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Όπως ζητήθηκε, κάθε χρόνο θα υιοθετούμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα, θα επισημαίνουμε τους τομείς προτεραιότητας, θα επισημαίνουμε τη, κατεπήγοντα όσον αφορά την έγκριση αυτών των εντολών και θα προσδιορίζουμε μαζί με τη βιομηχανία, θα παρουσιάζουμε όλα αυτά και στους ευρωπαϊκούς, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους τομείς κλειδιά στους οποίους πρέπει να εργαστούμε σε αυτόν τον τομέα. Πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές θα έχουμε την πρώτη ε, τελική έκδοση θα απορρεύσει αυτό και από μια διαδικασία συζήτηση με τα κράτη-μέλη και βάσει αυτού του κειμένου θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίηση θα λαμβάνουν υπόψη τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω το έχουν οριστεί από το πρόγραμμα εργασία. Αυτή είναι μια νέα σημαντική εξέλιξη για την τυποποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση θα ξεκινήσουμε και μια ανεξάρτητη αναθεώρηση του συστήματο τυποποίηση, ώστε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τον τρόπο λειτουργία του. Πιστεύω λοιπόν αυτή η τυποποίηση θα αποτελέσει φάκελο κλειδί. Αλλά πέραν αυτού του συγκεκριμένου εργαλείου τυποποίηση υπάρχουν δύο συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα ήθελα να ανακοινώσω σε αυτή την επιτροπή, επειδή είναι πολύ σημαντικά και τα παρακολουθείτε πολύ στενά. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για την εναρμόνιση των φορτιστών κινητών τηλεφώνων. Αυτό υποστηρίχθηκε στεναρά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή σα, Από τον κύριο Μάντρε ειδικότερα, αλλά και φυσικά από του καταναλωτέ, Πρόκειται για έναν τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και αρκετών δυσκολιών. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια θελοντική συμφωνία, αλλά τώρα αυτή η θελοντική συμφωνία που ήταν επιτυχής για αυτό το κοινό πρότυπο έχει λήξει από τα τέλη του 2012. Ζητήσαμε παράταση αυτής της συμφωνίας. Πρέπει να σας πω με λύπη μου ότι σημειώθηκαν διαφωνίες μεταξύ των υπογραφών των για παράταση αυτού του μνημονίου συνεννόησης. Και εμείς πραγματικά λυπούμαστε. Διότι οι καταναλωτές όλοι το είχαν θεωρήσει εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Εμείς παραμένουμε πεπισμένοι ότι οι καταναλωτές και οι κατασκευαστές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια παράταση αυτής της εναρμόνισης των φορτιστών και το ίδιο θα μπορούσε να συμβαίνει και για τις καινούργιες κατηγορίες κινητών τηλεφώνων, αλλά όχι μόνο για τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, ε, ταμπλέτες, όλες τις, ε, όλους τους τομείς. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω σε σχέση με αυτή τη συμφωνία ότι θα ε, παραγγείλει μια μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης. Εμείς εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα όπως μελλοντικές ε, εθελοντικές συμφωνίες, ενδεχομένως νομοθεσίες σε αυτό το τομέα. Όταν φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εθελοντικά πρότυπα, είμαστε υποχρεωμένοι να νομοθετήσουμε. Αυτό ήθελα να πω πολύ σαφώς και καθαρά ενώπιον αυτής της Επιτροπής. Υπάρχει και ένας δεύτερος τομέας, τα ηλεκτρικά οχήματα. Και εδώ συνεργαστήκαμε στενά με την Επιτροπή σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκατε αυτό το φάκελο. Είναι σημαντικό οι πρίζες, οι φορτιστές και τα ηλεκτρικά οχήματα να είναι διαλειτουργικά, να μην υπάρχουν διαφορές στις αγορές. Καταλήξαμε σε μια επιτυχία. Οι κατασκευαστές οχημάτων συμφώνησαν όσον αφορά την πρίζα εντός του οχήματος, αυτό συμφωνήθηκε και με τις Ηνωμένε Πολιτείε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι έτσι μπορούμε να έχουμε ένα παγκόσμιο πρότυπο, αλλά δεν σημειώθηκε επαρκής πρόοδος σε θέματα υποδομών. Ο κύριος Σταγιάννη έγραψε στους κατασκευαστές υποδομών και λόγω της απουσίας οποιασδήποτε πρόοδου σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να νομοθετήσει στη δέσμη μέτρων για τις υποδομές καυσίμων και αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει και την πρίζα τύπου 2 που θα εξοπλίζει την υποδομή που προορίζεται για το φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου τα εθελοντικά πρότυπα δεν έχουν λειτουργήσει και είμαστε υποχρεωμένοι να δράσουμε. Σα ενημερώνω λοιπόν ότι σήμερα ήδη η Κομισιόν υιοθέτησε αυτή την απόφαση. Τρίτο τομέα, στον οποίο θα ήθελα να αναφέρω, είναι κάποιε τομεακέ πρωτοβουλίε. Α ξεκινήσω από την αυτοκινητοβιομηχανία. Ξέρω ότι ενδιαφέρει ειδικότερα όχι μόνο όλου εσά, αλλά ειδικότερα και τον πρόεδρο. Οι εργασίες συνεχίζονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στην υποστήριξη της Επιτροπής σας. Η νομοθεσία της εσωτερικής ε, ε, αγοράς για μοτοσυκλέτες και τρακτέρ κατηγοριών Λάμδα και ΤΑΦ ε, επέτυχε. Αυτό, ενισχύθηκε αυτό μέσω των διατάξεων για την επιμέλεια των αγορών. Τώρα μπορεί να χρειαστεί επικαιροποίηση για έγκριση τύπου οχημάτων M, N και O. Αυτοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά και αυτή τη στιγμή ε, μπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι του CARS 21 που αποτελεί κομμάτι του σχεδίου CARS 2020 και χρειάζεται να βελτιώσουμε τις συνθήκες της αγοράς και την έξυπνη ρύθμιση. Ολοκληρώνουμε τον έλεγχο καταλληλότητα και θα καταλήξουμε σε κάποια πρόταση για αυτό το τομέα. Ένα δεύτερο τομέα που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη φετινή χρονιά είναι η αμυντική βιομηχανία στεναρή, ισχυρή βιομηχανική βάση στην αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανάπτυξη, θέσεων εργασία, καινοτομία, έρευνα. Είναι όμω κατακαιρματισμένο αυτό ο τομέα στην Ευρώπη. Εμεί, μετά βάσει των ειδηγιών του κυρίου Μπαρόσο, έχουμε μια task force που εργάζεται στην Κομισιόν και θα ακολουθήσει μια ανακοίνωση η οποία θα εγκριθεί μέσα στου επόμενου μήνε και που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την άμυνα επειδή το... Φέτος θα έχουμε μια, το 2013 θα έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Άμυνα και θα εστιαστούμε στη βιομηχανική πολιτική, την εσωτερική αγορά, την έρευνα και την καινοτομία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και κάποιες άλλες προτάσεις που έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί. Ο κανονισμός που απλοποιεί την ε, μεταβίβαση επιχανογέννητων οχημάτων αυτή η πρόταση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αναμένουμε με ανυπομονησία να συνεργαστούμε μαζί σας και με τον κύριο Μάντρης και τους κύριο εισηγητές για να ολοκληρώσουμε γρήγορα αυτό το φάκελο που αφορά την απλούστευση. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω την οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό. Αυτό είναι ένα από του ελάχιστου τομεί ε, υψηλή τεχνολογία, ε, τον οποίο ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να ενισχύσουμε το ρόλο μα και αναμένουμε να συνεργαστούμε στενά με την κυρία Βάλερ και τα άλλα μέλη για αυτή την πρόταση. Πριν ολοκληρώσω και ακούσω τι ερωτήσει σα, θα ήθελα να αγγίξουμε λίγο την εξωτερική δράση, διότι φέτο ε, θα είναι πολύ σημαντική η εξωτερική δράση και η Ευρώπη χρειάζεται, πρέπει να πω, ανοιχτέ αγορές. Σε εποχές έλλειψης ανάπτυξης, οι εταιρείε μας χρειάζεται να βγουν στο εξωτερικό, να διεθνοποιηθούν και να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε τρίτες χώρες. θα αντιστοιχεί αυτό σε 60-70% του ΑΕΠ το 2020 και σήμερα στην Ευρώπη μόνο μία από τις οκτώ εταιρείες βγαίνει εκτός χώρας και μία μόνο από τις τέσσερις εξάγει εκτός της εσωτερικής αγοράς. Αυτή η εξωτερική διάσταση λοιπόν είναι κρίσιμη σημασία. Όπως γνωρίζετε ο κ. Σταγιάννη ηγείται επιτυχώς τις αποστολές ε, ανάπτυξης σε συνεργασία με προεδρεύοντες εταιριών, με διάφορες εταιρείες πηγαίνουμε σε τρίτες χώρες και ενισχύουμε τα πρότυπα συνεργασίας, τη βιομηχανική πολιτική σε τομεί όπου είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδο. Αυτή τη στιγμή ο κ. Σταγιάννη βρίσκεται στο Περού με μια αντιπροσωπεία άνω των 40 εταιριών και στη Χιλή επίση, και θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωση με τις χώρες τη Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβική. Εγώ παρακολουθώ τις αποστολές του Ω Γενικό Διευθυντή και παρακολουθώ όλα αυτά και μαζί με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, και αυτό ήταν επιτυχέ και θα θέλαμε να σα αναφέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτή την Επιτροπή όσον αφορά τι επαγγελματικέ ευκαιρίε που ξαφνικά εμφανίζονται για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Φυσικά η ατζέντα του εμπορίου είναι πολύ σημαντική. Και φέτο, εκτό από τι διαπραγματεύσει με την Ιαπωνία, πολύ σημαντικό θέμα, έχουμε και την προοπτική διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένουμε την έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και ένας από τους τομείς κλειδί της διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, εφόσον υπάρξει κάποια σημαντική συμφωνία θα αφορά τα αριθμιστικά ζητήματα. Αυτό είναι ένα τομέα που μπορεί να γίνουν πολλά σε θέματα τυποποίηση, σύγκληση είναι εξαιρετικά περίπλοκο, δύσκολο, αλλά πολύ σημαντικό τομέα για τη διατλαντική διάσταση, διατλαντική διάσταση δεδομένου του όγκου του εμπορίου σε διατλαντικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας ότι η Επιτροπή σας ηγήθηκε της έγκρισης ε, νομοθετικών κειμένων πολύ σημαντικών όπως ε, τις οδηγίες για τις καθυστερημένες πληρωμές, ε, τα μηχανοκίνητα οχήματα, την κατασκευή, την τυποποίηση και στην τυποποίηση έχετε παίξει ρόλο κλειδί. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η υλοποίηση αυτών των φακέλων βρίσκεται σε εξέλιξη και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε γιατί εκτιμάμε ιδιαίτερα το εξαιρετικό σας έργο. Θα ήθελα όμως να πω επίσης ότι το 2013 θα χρειαστεί θα χρειαστούμε και κάτι πολύ σημαντικό που θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο στις 16 Μαρτίου η νέα οδηγία καθυστερημένων πληρωμών θα χρειαστεί να μεταφερθεί. Οι δημόσιες αρχές θα χρειαστεί να πληρώσουν τα χρέη τους εντός 30 ημερών. Και στην Ελλάδα και στις 27 χώρες μέλη. Θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να γίνει. Δεν γίνεται οι μικρομεσαίες μα επιχειρήσεις ως κομμάτι της αλυσίδας παραγωγής να δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε πιστώσει στον τραπεζικό τομέα και ταυτόχρονα να χρηματοδοτούν τις δημόσιες αρχές. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Αυτό το νομοθετικό κείμενο πρέπει να επιβληθεί. Ξεκινάμε μια ενημερωτική εκστρατεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η πρόταση προήλθε από αυτήν εδώ την Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να ζητήσουμε τη συμμετοχή σας και τη στήριξή σας σε μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Διότι χρειάζεται να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, χρειάζεται να ενημερώσουμε τον κόσμο. Διαφορετικά είναι σαν να μην έχουμε εγκρίνει καν αυτή την νομοθεσία και αυτή η νομοθεσία έχει εγκριθεί από όλα τα κράτη-μέλη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να μεταφερθεί. Και αν σε μερικέ χώρε ε, είναι δυνατή η πληρωμή εντό των προθεσμιών, δεν ξέρω για ποιο λόγο να μην το κάνουμε. Θα χρειαστεί λοιπόν να επιμείνουμε επ' αυτού και θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας. Εγώ προσωπικά είμαι ανυπόμονος να συνεργαστώ στενά με την Επιτροπή σας όταν η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώνουν δυνάμεις μπορούμε να είμαστε αίτητοι. Ευχαριστώ πολύ. Well, Πρόεδρος, νομίζω ότι μιλώ εκ μέρου όλων των μελών της Επιτροπής λέγοντας ότι πραγματικά αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα την ποιότητα των επαφών που είχαμε με τη Γενική Διεύθυνση Enterprise όχι μόνο σε σχέση με, θέματα της εσωτερικής αγοράς. Όταν ήρθε πέρσι ο αρμόδιος επίτροπος εδώ και είπαμε ότι θέλουμε να ξαναδούμε ορισμένα πράγματα για τα εμπορεύματα και τα λοιπά, ε, έτεινε το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών που αναφέρατε. Ήταν ένα άλλο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρε ιδιαίτερα. Λοιπόν, ε, βλέπω ότι αρκετοί ζητούν το λόγο, τέσσερις-πέντε τουλάχιστον. Ας αρχίσουμε με τον κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κρέσπο για τα, την παρουσίαση που μας έκανε. Ας ξεκινήσουμε τις πληρωμές. Άκουσα από τον κλάδο ότι δεν παραδίδουν φάρμακα στην Ελλάδα γιατί ε, για να πάρουν τα χρήματα πρέπει να περιμένουν τρία χρόνια και μετά από τρία χρόνια αρχίζουν διαπραγματεύσεις για εκπτώσεις στα φάρμακα τα οποία έχουν ήδη παραδοθεί μιλάμε για τρία χρόνια στην Ελλάδα, ένα χρόνο στη Ρουμανία. Να περάσουμε από αυτά τα χρονικά διαστήματα στις 30 μέρες μου φαίνεται τεράστιο πράγμα. Ε, μακάρι να μπορέσει η Κομισιόν να το κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι αυτό που είπατε για την ε, επανεκβιομηχάνηση ορισμένων της Ευρώπης ε. στη Γερμανία βλέπουμε ότι ε, σε ορισμένους κλάδους είμαστε πολύ κοντά στο 1 τρίτο του ΑΕΠ έτσι στην Αγγλία στη μεγάλη ε, Βρετανία ε, τα πράγματα ήταν, ξεκίνησαν από το 10% και έχουν αυξηθεί. Στη Γαλλία υπάρχουν αντίστοιχα νούμερα. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολος ο γενικός αυτός στόχος που θέσατε. Έτσι. Παλιά βέβαια, αλλά ε, τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη ερχόντουσαν από την Αγγλία. Αλλά ε, όμως και τώρα έρχονται πολλά αυτοκίνητα από την Αγγλία απλώ δεν ανήκουν σε βρετανικέ εταιρείε. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να δούμε πώ μα ενδιαφέρει να ε, προχωρήσουν τα πράγματα. Ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε το ITS. Ε, υπάρχει θέμα Υπάρχει και θέμα τιμών, ε, γιατί γίνονται ορισμένα πράγματα τα οποία βαίνουν αντίθετα προς την ε, πάνεκ στην οποία αναφερθήκατε. Τώρα, για το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων. Όπως ξέρει ο Μάλκον, κάναμε ορισμένα πράγματα, πήραμε κάποιες αποφάσεις και ζητήσαμε να εφαρμοστούν σε 6 μήνες. Και μετά το Συμβούλιο, δηλαδή οι χώρες μέλη, μας είπαν όχι σε 6 μήνες, αλλά πρώτη-πρώτη του 2014. Τα τελωνία, γιατί μιλάμε για ε, εποπτεία της αγοράς ή θέματα ασφάλειας που ελέγχονται από τα τελωνία. Τα τελωνία όμως είναι, ε, δεν έχουν επαρκές προσωπικό Πώς λοιπόν μπορούμε να προωθήσουμε τα πράγματα έτσι όπως θέλουμε και να αναθέσουμε περισσότερους ελέγχους στα ε, τελωνία ε, όταν τα κράτη-μέλη δεν έχουν, βάζουν αρκετό κόσμο στα τελωνία. Έρχομαι τώρα στην τυποποίηση. Τα ε, γίνονται συνεχώς με μεγάλες αλλαγές στην αγορά. Τα πράγματα είναι ρευστά. Εσείς λέτε τώρα ότι αν δεν υπάρξουν εθελοντικές συμφωνίες τότε θα νομοθετήσετε. Εγώ θα έλεγα πιέστε ακόμη περισσότερο για εθελοντικές συμφωνίες διότι διαφορετικά η οποιαδήποτε νομοθεσία στην οποιαδήποτε νομοθετική σας δράση θα σας ξεπεράσει η πραγματικότητα. Αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα. Ε. Είναι όλα αυτά που είπατε, είναι πράγματα που πράγματα θα βοηθήσουν στη βελτίωση τη εσωτερική αγορά. Θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη, θα βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων ε, απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο κύριος Χάτσισον ο επόμενο ομιλητή και μετά θα απαντήσει ο κύριος Καλέχα. Χάτσισον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την παρουσίαση είναι παράξενο που δεν έχουμε περιορισμό στο χρόνο μιλίας. Έχουμε χρόνο ε, για να κάνουμε ερωτήσεις και να πάρουμε απαντήσεις. Αυτό είναι πολύ καλό το χαιρετίζω. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση μα ιδιαίτερα τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πριν από μερικά χρόνια όταν πρώτο ήρθα εδώ αυτό δεν ήταν τόσο προφανές. οι ψηφοφόροι μου τουλάχιστον συνεχίζουν να απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε όμως ότι ε, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και ε, ίσως αρχίσουν να περικόπτουν ε, αν δεν το έχουν κάνει ήδη θέσεις εργασίας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να τις βοηθήσουμε και όσον αφορά την απλούστευση και όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Τελικά είναι και λίγο παράξενο να μιλούμε για απλούστευση όταν βλέπουμε εδώ τόνους χαρτιού που σχετίζεται ας πούμε με, τις, ε, ε, νομο, με την νομοθεσία για τις προμήθειες ε, και τη γραφειοκρατία που επεμβαίνει στις προμήθειες. Ε, χρειάζεται πραγματική απλούστευση για, τις μικρο, για τη μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορεί να υποβάλει κάποια προσφορά, να εκδηλώσει ενδιαφέρον να υποβάλει με κάποια προσφορά και να λάβει μέρος κάποιο διαγωνισμό ε, για να κερδίσει κάποια συμβόλαια. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κατά πόσον πιστεύετε ότι θα μπορούς να μας πείτε αν θα μπορούσαν να γίνουν αν θέλετε κάποιες εξαιρέσεις ή ξέρω εγώ απλουστεύσεις για τις δημόσιες ε, προμήθειες να μοριοδοτούνται τρόπον την η εντοπιότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή κάτι τέτοιο δεν ξέρω για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα για τις καθυστερημένες πληρωμές χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αν υπάρχει, δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα α, για τις μικρομεσαία επιχείρηση για τον οποιοδήποτε επιχειρηματία τελικά να έχει κάνει αντιμε... την υποχρέωσή του να έχει παραδώσει το εμπόρευμα και να μην πληρώνεται. Αυτό είναι πρόβλημα και στην ε, Σκοτία είναι πρόβλημα. Βεβαίω, ευτυχώ, οι δημόσιοι φορεί στη Σκοτία έχουν κάνει αρκετές προσπάθειες ε, αλλά οτιδήποτε γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι καλό. Τέλος, για την εξωτερική πτυχή στην οποία αναφερθήκατε, μπορείτε να μας πείτε σε ποιο βαθμό η Κομισιόν μπορεί να εξασφαλίσει ότι όταν γίνεται, ας πούμε, μια εμπορική συμφωνία μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το εισαγόμενο, το πούμε, προϊόν ανταποκρίνεται στις ε, προδιαγραφές ή στις απαιτήσεις που έχουμε εμείς στο εσωτερικό μας ή στην, στην περιοχή μας. Είναι ε, σημαντικό αυτό νομίζω. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για το νούμερο ένα προϊόν εξαγωγής της Σκωτίας που είναι το whisky. Ε, ε, το whisky πρέπει να ιδιαίτερα αυτό που αποστάζεται στην ε, ε Σκοτία είναι πάρα πολύ καλό για την ανθρώπινη υγεία όταν βέβαια δεν γίνεται κατάχρηση αυτού. Λοιπόν, μπας περιπτώσει επειδή και άλλοι προσπαθούν να παράγουν ουίσκι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε τι γίνεται με τις διεθνείς ε, εμπορικές συμφωνίες. Ειδικά για το ουίσκι είναι πολύ σημαντικές οι συμφωνίες αυτές. Πρόεδρος, ο μια χαρά μου φαίνεται ε, και ξέρω ότι πίνει σκοτσέζικο ουίσκι, βέβαια με τριοπαθός, ε. Λοιπόν... So, like to... Θα ήθελα να δώσω κάποιες απαντήσεις. Πρώτα, για τις ερωτήσεις που έγινε. Λοιπόν, για τον κύριο Κρόιτσμαν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη δουλειά που κάνετε στο πρόγραμμα COSME που είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει αποκλειστικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο θα στηρίξει οικονομικό και σε με, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ε, θα υποστηρίξει γυναίκες, νέους επιχειρηματίες θα ε, ε, βοηθήσει στη μείωση της γραφειοκρατίας και τα λοιπά. Αυτό το πρόγραμμα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε να στεφθεί με επιτυχία το πρόγραμμα αυτό. Θα το δούμε αργότερα βεβαίως αυτό, αλλά ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Κρόιτσμαν που έχει αναλάβει ηγετική θέση για το πρόγραμμα αυτό. Για τι καθυστερημένε καθυστερημένες Ο μέσος όρος καθυστερήσεων στη, μεταξύ των 27 χωρών δεν είναι τρία χρόνια βεβαίως. Ο μέσος όρος είναι 183 μέρες. Ε, ο σκοπός μας, ο στόχος μας είναι 30 μέρες που είναι μεγάλη μείωση από τις 183 έτσι λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό και μαζί με το Κοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι τα κράτη-μέλη, οι δημόσιοι φορείς υποστήριξαν, συνυπέγραψαν το νομοθετική, τις σχετικές νομοθετικές πράξεις. Το δέχτηκαν δηλαδή. Να πούμε κιόλας ότι πρέπει να υπάρχουν πρακτικές και θα πρέπει να μιμηθεί κανεί αυτές τις βέλτικες πρακτικές. Γιατί κάποιες χώρες τα καταφέρνουν και κάποιες άλλες όχι. Ας αντιγράψουμε αυτές τις χώρες που, που τα καταφέρνουν. Θέλουμε επίσης να κάνουμε ένα διάλογο με εκείνες τις χώρες που έχουν προβλήματα Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η κατάσταση. Διαφορετικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας είναι καταδικασμένες. Και γι' αυτό η δική σας συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλες εσείς από τις σε όλες τις χώρες θα πρέπει να εξηγήσετε τα πράγματα. Εάν καταφέρουμε να περάσουμε νομοθετικές διατάξεις εδώ και να τηρούνται τότε σώζουμε τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις γιατί πολλές από αυτές καταστρέφονται επειδή ακριβώ δεν μπορούν να εισπράξουν τελικά. Πρέπει λοιπόν να πετύχει αυτό το ε, να πετύχει αυτή η προσπάθεια. Τώρα, για την ανάπτυξη και την επανεκβιομηχάνηση. Ε, αναφερθήκατε σε αυτό και είπατε ότι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν προκλήσεις. Ε, η κυρία Μέρκελ αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπε ε, 7% του πληθυσμού της γης, 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και 50% των κοινωνικών δαπανών του κόσμου και υπάρχουν και προβλήματα ανταγωνιστικότητα. Και εγώ θα έλεγα και πιστεύω πληρώνουμε και τις πιο, α, την πιο ακριβή ενέργεια, τις ψηλότερες τιμές για ενέργεια στον κόσμο. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και εδώ. Και υπάρχει και φοβερός διοικητικός φόρτος, κανονιστικός φόρτος αν θέλετε, για τις επιχειρήσεις μας. Κάπως λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, των οποίων την πολυπλοκότητα δεν υποτιμούμε βεβαίως, αν καταφέρουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, θα θα τα καταφέρουμε. Προσπαθούμε Παρακολουθούμε το πώς προχωρούμε. Ξέρουμε ότι η κατάσταση με των διαφορών χωρών είναι ανισομέρειες. Δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τις δεξιότητες, τις ειδικότητε. Οι χώρες στις οποίες οι επιχειρηματικότητα συνδέεται περισσότερο με την παιδεία. Εκεί ο κλάδος των επιχειρήσεων με την παιδεία, εκεί τα πράγματα πάνε καλύτερα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη στις ιδιαιτερότητες αυτές, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες για να μπορέσουμε με έναν έξυπνο τρόπο να επιτύχουμε μια συνεπή επανεκβιομηχάνηση. Τώρα, για την ασφάλεια των ε, προϊόντων που είπατε. Εδώ και εδώ υπάρχει σοβαρό, σοβαρή πρόκληση, διότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέσουν τους πόρους. Ε, να φροντίσουν, να ελέγχουν και αυτά όπως είπε ο κύριος Χάτσον προηγούμενα. Ε, Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένα προϊόν που έρχεται από μια τρίτη χώρα ανταποκρίνεται στις απαιτήσει που έχουμε εμείς στο εσωτερικό μας. Εδώ μπορούμε να έχουμε νομοθετικές διατάξεις και κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά πρέπει να τις ελέγχουμε κιόλας. Πριν από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς ήμουνα στο, στην Κίνα. Κάναμε έναν τον παραδοσιακό διάλογο με τους ε, Κινέζους και συζητήσαμε Υπάρχουν βεβαίως και προγράμματα κατάρτισης ε, τα οποία ε, μέσω των οποίων ε, εκπαιδεύουμε αυτούς οι οποίοι έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν ότι την συμμόρφωση των εισαγωγών από την Κίνα. Και οι Κινέζοι ενδιαφέρονται όμως τα προϊόντα τους να είναι σύμμορφα. Εκείνο όμως επίσης που κάναμε είναι ε, κάναμε μία ολόκληρη δουλειά για τις προδιαγραφές και την τυποποίηση να είναι και στα αγγλικά και στα κινέζικα ε, και να είναι υποχρεωτικό αυτό τουλάχιστον για το μηχανικά προϊόντα έτσι ούτω ώστε να ξέρουν και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει συμμόρφωση. Και αν δεν υπάρχει συμμόρφωση τότε πρέπει να πάρουμε τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται ε, ούτως ή άλλως από την νομοθεσία. Τώρα, για τα, την τυποποίηση, εδώ η βιομηχανία πρέπει να δράσει τα πρότυπα, δεν είναι νομοθεσία. Αλλά εάν τελικά αναγκαστούμε να καταφύγουμε στην νομοθεσία. Αν δηλαδή οι βιομηχανίες δεν αυτορυθμίζονται ή δεν ε, λύνεται το πρόβλημα των προτύπων από την ίδια τη βιομηχανία, τότε σαν τελευταίο καταφύγιο μπορεί να προσφύγουμε στην νομοθετική ρύθμιση. Είπατε στο τέλος παρέμβασή σας ότι ε, αν γίνουν όλα αυτά πραγματικά θα βελτιωθεί, ε, θα μιλάμε για βελτίωση εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χάτσον μίλησε για τις προκλήσεις των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι, και ε, στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχει πολύ προσωπικό που και υπάρχουν και οι άνθρωποι ειδικοί που μπορούν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τις οποίες έρχομαι σε επαφή μου λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να πουλήσουμε προϊόντα διότι ε, ε κατακλυζόμεθα από έγγραφα, από γραφειοκρατία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, τοπικό επίπεδο, ε, περιφερειακό επίπεδο και ευρωπαϊκό <laughs> επίπεδο. Ορίστε τα χαρτιά ντάνε ολόκληρας. Εγώ είπα ναι, μπορώ να βοηθήσω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι πραγματικά πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απλούστευση. Η, αυτή η διαβούλευση για τις, τα 10 καλύτερα του top 10 που λέγαμε προηγούμενα ε, θα βοηθήσει ε, μας ενδιαφέρει η έξυπνη νομοθεσία, μας ενδιαφέρουν, η, ε, ενδιαφέρει η απλούστευση των τεστ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να και το σωρευτικό αποτέλεσμα της νομοθεσία θα πρέπει να δούμε διότι καμιά φορά εκείνο που ενοχλεί δεν είναι η επιμέρους κανονιστική ρύθμιση αλλά η σώρευση πολλών τέτοιων ρυθμίσεων που δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού τελικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα για τις δημόσιες προμήθειες που μιλήσατε. Κοιτάξτε, 17 τα 100 του ευρωπαϊκού ΑΕΠ είναι οι δημόσιες ε, προμήθειες. Μόνο ένα τρίτο αυτό πάνε πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι προσπαθήσαμε κάτι να κάνουμε για αυτές. Έτσι, είπαμε ότι μπορεί κανείς να μειώσει το συνολικό ποσό, ε, ε αν μπορούμε να έχουμε μειώσουμε για μεγάλες προμήθειες το ποσό, να κατακαιρματίσουμε αν θέλετε το ποσό, τότε μπορούν να συμμετάσχουν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που μας ενδιαφέρει επίσης είναι οι ηλεκτρονικές προσφορές και αυτό θα, θα βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό το είδαμε να γίνει στις ορισμένες χώρες. Τρίτη δυνατότητα, αν κερδίσει η προσφορά σας, τότε θα πρέπει να υποβάλλετε όλα τα δικαιολογητικά στο τέλος ο υπερθεματιστής να πρέπει να το κάνει αυτό αλλά μην το βάζετε από την αρχή είπαμε ούτω διότι ουσιαστικά είναι αποτρεπτικό στοιχείο για τη μικρομεσαία επιχείρηση όχι Βάλτε την υποβολή δικαιολογητικών και τα λοιπά στο τέλος, σε αυτόν που, του οποίου προσφορά κέρδισε. Αυτό βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι τι άλλο που είπατε, διεθνείς διαπραγματεύσεις, διεθνείς συμφωνίες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Βεβαίω όλο και περισσότερα εστιάζουμε στα κανονιστικά θέματα με τις τρίτες χώρες, με την Ιαπωνία, δεν ξέρω, με και τα λοιπά. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να διαπραγματεύεται, αλλά και εμείς ε, ε, συμμετέχουμε με μια έννοια και βεβαίω εκείνο το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η προστασία τη καταγωγής. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι και για το σκοτσέζικο ουίσκι και για το κρασί ριόχα που είναι το δικό μου το ποτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την ποιότητα των προϊόντων να ε, ελέγχεται ε, η καταγωγή να αποφύγει η κυκλοφορία προϊόντων ε, που δεν είναι πραγματικά ε, τα προϊόντα τα οποία περιμένουμε. Και πριν να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ζητούμε να γίνει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ποια, ε, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις, τι πρέπει να τσεκάρουμε, τι πρέπει να ελέγχουμε για να είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και τα βασικά μας συμφέροντα θα προστατευθούν. Σας διαβεβαιώ ότι το κάνουμε αυτό, αλλά βεβαίως για πιο ειδικά θέματα θα ξακουβεντιάσουμε τα θέματα. Ναι. Ξέρω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Η κυρία Σάλοβα και η κυρία Κολελάγκα. Κυρία Σάλοβα πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ, με τη σειρά μου, θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας. Και έχω παρακαλώ μία συγκεκριμένη ερώτηση για τις μεταφορές. Αναφερθήκατε σε κάποιες δραστηριότητες, αλλά για μένα λείπει μία από αυτά που είπατε. Και αυτό είναι το σύστημα e που έχει να κάνει με τα ατυχήματα και πώς δηλαδή κάποιος όταν έχει ατύχημα μπορεί να ενημερώσει ηλεκτρονικά τις ε, αρμόδιες αρχές είναι κάτι που ψηφίσαμε εμείς θετικά με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Οπότε από το 2015 θα είναι υποχρεωτικό ένα τέτοιο σύστημα, αλλά για να εφαρμοστεί χρειαζόμαστε μια πρόταση κανονισμού από εσάς Για να δούμε σε ποιο σημείο ακριβώς του πίνακα πλεύσης, του οχήματος τέλος πάντων, θα βρίσκεται ο μηχανισμός αυτός. Ο κύριος Κοχ, που είναι ο συγκητής μας ε, από την Αρμόδια Επιτροπή, ήρθε σε επαφή με τον κύριο Ταγιάννη, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι μπορούμε να περιμένουμε φέτος κάποια αποτελέσματα από αυτού. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε εσείς. Έπειτα το φθινόπωρο που μας πέρασε πήγα στο Ζάγκρεπ σε μια διάσκεψη όπου ήταν παράγοντες από διάφορες χώρες και από χώρες όπου γίνονται δοκιμές ήδη για το σύστημα αυτό. Εκεί λοιπόν συναντήθηκα και με τους εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας που λένε ότι και εκείνοι περιμένουν την πρόταση κανονισμού για να μπορούν να έχουν κάποια βεβαιότητα, να ξέρουν τι να περιμένουν, τι, τι προσαρμογές πρέπει να κάνουν και αυτοί. Φυσικά και είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε ασφάλεια, κανένας δεν το αμφισβητεί. Αλλά ο κόσμος χρειάζεται κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για να έχει βεβαιότητες. Ευχαριστώ για την απάντησή σας εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Κυρία Κονελίνη. Ευχαριστώ πολύ πρώτα πρώτα για την παρουσίασή σας και Χαίρομαι ιδιαίτερα που τονίσατε δύο πράγματα. Από τη μια μεριά τη διοικητική απλούστευση, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ισχύει και για την τοπική αυτοδιοίκηση στη Γερμανία, γιατί ήμουνα εγώ μέλος της τοπικής αποδιοίκησης αυτοδιοίκηση και ξέρω πολύ καλά ότι ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε όλη τη γραφειοκρατία η οποία ε, απαιτεί το. Επίσης χαιρετίζω τις 30 μέρες που θέσατε σαν στόχο για τις ε, ε καθυστερημένες ε, πληρωμές. Ε, βεβαίως μπορεί να ισχύει αυτό για, πάλι για ορισμένους φορείς τοπικής αυτοδίκησης, αλλά τελικά κατέληξε σπορ. Ε, Πραγματικά ε, πολλοί φορείς δεν πλήρωναν έτσι γιατί δεν ήθελαν να πληρώσουν. Βέβαια στα τρία χρόνια είναι υπερβολικά πολύ. Από εκεί και πέρα η, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κρόιτσμαν ε, ότι γιατί Εάν τελικά η, η βιομηχανία δεν αυτορυθμιστεί ή δεν υπάρχουν εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων κλάδων και των διαφόρων χωρών, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτή την περίπτωση τον καταναλωτή ή τον πολίτη της Ευρώπης. Και εκεί θα πρέπει να καταφύγουμε πλέον στη τελευταία, ε, στο, τελευταίο μέτρο που έχουμε στη διάθεσή μας να νομοθετήσουμε διότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται ορισμένα πράγματα. Thank you very much. First of all, I would like... Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σανάλοβα, πρώτα απ' όλα, που επιστήνει την προσοχή μου στο σύστημα αυτό e-call, ηλεκτρονική κλίση δηλαδή. Όντω, δεν κάλυψα στην παρουσίασή μου όλα τα θέματα, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στο τεχνικό σκέλος και είναι σημαντικό γιατί είναι μια πολύ δυνατή διάσταση αυτή η τεχνική. Σας ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθείτε τόσο στενά αυτό το ζήτημα. Όλα τα νέα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν αυτό το σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης. Και ο λόγος είναι ότι θέλουμε να μειώσουμε τα μοιραία ατυχήματα στο δρόμο. Το χρονικό διάστημα δηλαδή που θα μεσολαβεί από το ατύχημα μέχρι την ε, βοήθεια μειώνεται πάρα πολύ μέχρι να φτάσει η βοήθεια. Σας επιβεβαιώνω λοιπόν ότι όντως έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος και ότι θα είναι μια πρόταση αυτή η οποία θα έρθει σύντομα γιατί είναι σημαντικό θέμα, το εξετάζουμε έχω παρακολουθήσει όλες τις πρωτοβουλίες και σας διαβεβαιώνω, περιλαμβάνεται και αυτή. Θα υποβάλουμε στον κύριο Ταγιάννη βέβαια το σχέδιο και θα είναι μια τελική πρόταση προς εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ που μου το θυμήσατε. Έρχομαι τώρα στην κυρία Κόλλη Λάγκεν. Και αυτό που είπατε για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές. Είναι θλιβερό που υπάρχουν τέτοιες κακές πληρωμές, ότι δηλαδή κάποιες δημόσιες αρχές λένε εγώ δεσμεύομαι, αλλά μετά δεν σέβομαι, δεν τηρώ τις προθεσμίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονται και μου λένε μερικέ φορές, ξέρετε τι μας συμβαίνει εμά αν δεν πληρώσουμε τους φόρους μας ή αν δεν πληρώσουμε τα χρέη μας στη δημόσια διοίκηση. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι δίκαιο. Οι οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητούν σε ορισμένε χώρες αποζημιώσεις από το κράτος. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Αλλά για να αλλάξουμε την νοοτροπία πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, όλες οι πλευρές. Η κοινή γνώμη πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό πιστεύω ότι εσείς έχετε να παίξετε σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ο κύριος Σταγιάννη θέλει αυτή την εκστρατεία φέτος. Έχουμε προχωρήσει πολύ. Ορισμένε χώρες πρέπει να ξέρετε ότι το αντιλαμβάνονται ήδη. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα, γιατί η οδηγία αυτή είναι επαναστατική. Έχει να κάνει με όλους τους τομείς. Υπάρχει και η προθεσμία των 60 ημερών για τις πληρωμές μεταξύ ατόμων με κάποιες εξαιρέσεις. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο αυτό. Και όπως λέτε κι εσείς, πρέπει να τηρηθεί η προθεσμία και να συνεργαστούμε έτσι ώστε τα στο τέλος να έχουμε ομοιόμορφους κανόνες που να ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντήσατε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις πλήρως και χαίρομαι που αναγνωρίζετε και εσείς τη δικιά μας τη δουλειά. Γιατί όντως και εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια συνέχεια στην νομοθεσία που αποφασίζουμε. Για το θέμα δεν είναι μόνο να την εξετάζουμε και να την αποφασίζουμε, πρέπει να βλέπουμε και πώς προχωράει, ότι γίνεται πραγματικότητα. Υπάρχουν και πρωτοβουλίες που παίρνει το Κοινοβούλιο. Σίγουρα στην ημερήσια διάταξη θα υπάρξουν και θέματα για την τυποποίηση ακόμα και οι σχετικές οργανώσεις κάνουν πολλή δουλειά σε αυτό το θέμα. Εγώ με την έτσι συναντήθηκα χτες με τις εκπροσώπους της ΕΝΕΛΕΚ. Είναι ε, πολύ σημαντικό θέμα η τυποποίηση και έχει βέβαια και διεθνή διάσταση. Πολύ χάρηκα πάντως που στην αρχή αναφερθήκατε στην οδηγία 9834. Όπως είπατε, είναι μια σημαντική οδηγία αυτή προκειμένου να λειτουργήσει καλά η ενιαία αγορά. Ο κύριος Τάκμα, που είναι ένας από τους κύριους ερευνητές σε αυτό το θέμα, δημοσίευσε ένα βιβλίο που μιλάει για την θέση ισχύ της ενιαίας αγοράς και λέει ότι το βασικό είναι να υπάρχουν τα σωστά εργαλεία. Ίσως λοιπόν ασχοληθούμε με τους συντονιστές για να κάνουμε κάτι όσον αφορά την εφαρμογή σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ο Κάρλο Βατινέλη βλέπω ότι είναι εδώ, που έχει συνεργαστεί μαζί μας για πολλά ζητήματα. Λοιπόν, θα μεταφέρετε στον κύριο Ταγιάννη αυτά που είπαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στη χρονιά, ώστε να πάρουμε τις προτάσεις σας έγκαιρα, εκεί που μας τις υποσχεθήκατε. Με το συνηθισμένο μας τρόπο θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα διάφορα ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε πάλι. Στο επανειδήνιο. So, if we uh, now Τώρα, περνάμε στα δύο τελευταία θέματα που έχουμε να εξετάσουμε ακόμα σήμερα. Πρώτα, για όσους μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο. Ή και σε εσά να το πω ότι σχετικά με τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι οι κύριοι σκιώδεις συζητητές δεν ήταν εδώ σήμερα, έχει σαν αποτέλεσμα Ashley Fox ζήτησε να το αναβάλουμε το θέμα αυτό για το Φεβρουάριο. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι συνεχίζεται η δουλειά, έτσι. Όσοι δηλαδή μας παρακολουθούν να ξέρουν ότι αν έχουν σχόλια ευχαρίστως να τα στείλουν στην Ashley Fox. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα. Θα ασχοληθούμε με δύο σημαντικές γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής μας. Για να δώσουμε τα φώτα μας και εμείς, μια που είμαστε η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά. Πρώτα απ' όλα, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θα δώσουμε τα φώτα μας, τη γνωμοδότησή μας δηλαδή, για το περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των μουλκόμενών τους, που είναι το σημείο 20 που είναι δικό μου και το άλλο θέμα είναι κλινικέ δοκιμέ φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάρρευση τη οδηγία 2001 2001-20 του Κριστιαν Σιλβίου Μπουσόη. Η κυρία Λεγκρίπ θα μιλήσει όμως εκ μέρους του κυρίου Μπουσό, έτσι δεν είναι. Δεν βλέπω άλλους σκιώδεις. Η κυρία Σαντεμόσε δεν είναι από τους σοσιαλιστές, ούτε άλλοι. Τέλος πάντων, θα αρχίσει όμως η διαδικασία παρόλα αυτά. Επίσης, για να ελέγξω, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Ωραία. Μας παρακολουθείτε. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής. Ο κύριος Ρης. Καλώς. Άντριου Ρης. Ωραία. Θα σας δώσω μετά το λόγο. Πρώτα να ακούσουμε την παρουσίαση από τον Κρίστιαν Σιλβίου Μπουσόη. Ευχαριστώ. Είναι η πρώτη συζήτηση αυτή που έχουμε και θα έχουμε και άλλη φορά την ευκαιρία, πόσο ξέρω, να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε συζητήσει πολύ με τους σκιώδες εισηγητές, οι οποίοι έχουν ετοιμάσει τροπολογίες για την βελτίωση της οδηγία αυτής. Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική νομοθεσία γιατί θέλει να διευκολύνει την πρόσβαση στην εναλλακτική και νέα ιατρική από πλευρά των καταναλωτών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ότι τέτοιες ε, μέθοδοι και πρακτικές εγκρίνονται να καλύπτονται και από την ασφάλιση. Την τελευταία φορά το Κοινοβούλιο που συζήτησε για τον ορίζοντα 2020 συζητήσαμε για την οδηγία διαφάνειας. Τώρα θέλουμε να ενισχύσουμε ε, τα πράγματα και να περάσουμε και στις κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Και πρέπει να σας πω ότι η οδηγία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας δεν έχει πετύχει τους στόχους της. Και μάλιστα ορισμένοι συνάδελφοι θεωρούν ότι η οδηγία αυτή είναι υπεύθυνη για το 25% μείωση των κλινικών δοκιμών που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 μέχρι το 2011 ότι το σημερινό σύστημα δεν είναι ικανοποιητικό για τις δοκιμές και μειώνουν, όπως είπαμε, τις κλινικές διακοπές, δοκιμές που είναι πολύ σημαντικές. Το θέμα είναι να απλοποιηθεί τώρα το σύστημα, να γίνει πιο αποτελεσματικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ελκυστική για κλινικές δοκιμές και για κλινικές έρευνες γενικότερα. Συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έκανε. Ξέρω ότι υπήρξε ευρεία διαβούλευση ε, επί του νομοθετήματος αυτού με το κοινό και αυτό φαίνεται στην πρόταση. Πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από τους διάφορους φορείς με τους οποίους μίλησα μέχρι τώρα εκφράσουν την ικανοποίησή τους από την πρόταση αυτή. Περιλαμβάνει λίγες τροπολογίες πρέπει να σας πω, προκειμένου να διευκρινιστούν κάποιες πτυχές που δεν αλλάζουν όμως τον προσανατολισμό που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο νομοθέτημα αυτό. Το θετικό είναι ότι πρόκειται για κανονισμό πια. Νομίζω ότι έτσι ομοιόμορφα θα τεθεί σε εφαρμογή και αυτό είναι προτιμότερο. Τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ λιγάκι σε 6-7 πτυχές που θεωρώ ότι είναι σημαντικές και θα σας πω μετά ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Πρώτον, για το πόρταλ, την δικτυακή πύλη. Θέλουμε μια αποκεντρωμένη διαδικασία. θα έχει δυσκολίε, ακόμα και αν είναι ιδανική. Γι' αυτό προτιμάω αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να φτιάξει μια ενιαία δηλαδή δικτυακή πύλη για τι κλινικέ δοκιμέ. Είναι ένα καλό συμβιβασμό και είναι ό,τι καλύτερο στη σημερινή κατάσταση, γιατί έτσι θα απλοποιηθεί η διαδικασία αιτήσεων και θα διευκολύνει τις πολυεθνικές κλινικές δοκιμές. Τώρα, για το σημείο 1 και 2. Προτείνει να χωριστεί η εξολόγηση σε δύο τμήματα. Στο ένα τμήμα που συνεργάζονται οι χώρες μέλη και καλύπτονται εκεί θέματα για τα οποία μπορούμε να έχουμε μια κοινή αξιολόγηση, όπως είναι θεραπευτικά ωφέλη, κίνδυνοι για τον ασθενή κλπ. Και ένα δεύτερο τμήμα το οποίο καλύπτει πράγματα τα οποία είναι πιο πολύ σε εθνικό επίπεδο και κάθε χώρα χωριστά θα τα κάνει μόνη της. Είναι όμως σημαντικό εδώ να διευκρινίσουμε ότι ενώ η τελική απόφαση καλύπτει και τα σημεία 1 και 2, οι κλινικές δοκιμές μπορούν να αρχίσουν χωρίς καθυστερήσεις λόγω άλλων ε, εκτιμήσεων αξιολογήσεων που να χρειάζονται. Τώρα το θέμα της ηθικής διάστασης που αναφέρεται στο κείμενο. Δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας. Γι' αυτό ακόμα και αν αναφέρεται ρητά, εγώ προτείνω ένα νέο άρθρο για να διευκρινιστεί ότι η αξιολόγηση των τμήματων 1 και 2 καλύπτει και τις ηθικές πτυχές. Αναφέρεται και οι ηθικές επιτροπές, όμως δεν έχουν τις ίδιες δομές οι χώρες μέλη και σε μερικές περιπτώσεις δεν ονομάζονται καν επιτροπές ηθικής και μερικές φορές είναι και σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι σε εθνικό. Οπότε αφήσουμε τις χώρες μέλη να οργανώνονται όπως θέλουν όσον αφορά την ηθική αξιολόγηση. Μόνο που αυτή πρέπει να γίνεται μέσα στις προθεσμίες. Χρονοδιαγράμματα τώρα για τις δοκιμές. Πρέπει να δούμε τι δυνατότητε έχουν τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν κλινικέ δοκιμέ σύντομα. Με το τρέχον σύστημα Χρειάζεται περισσότερο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο, προκειμένου να δίνεται άδεια για κλινικές δοκιμές. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Καναδά για παράδειγμα, είναι πιο γρήγορα εκεί τα πράγματα. Γι' αυτό ε, με τον κανονισμό αυτό προσπαθούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να μπορούν έτσι ομαλά να παίρνουν αποφάσεις. Ελαστικότητα. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να προσφέρει κάποια ελαστικότητα και χαίρομαι για το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα να προστίθεται μια χώρα στις πολυεθνικές κλινικές δοκιμέ. Βέβαια, δεν είναι σαφές από το κείμενο πότε μπορεί να γίνει το αίτημα αυτό επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, νομίζω ότι πρέπει μέσα στο σύστημα να συμπεριλάβουμε το ότι μπορεί να υποβληθεί τέτοιο αίτημα για νέα χώρα μέλος, μόνο εφόσον όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν κοινοποιήσει την απόφασή τους για την αρχική αίτηση. Επιπλέον πιστεύω ότι πρέπει να αποσαφανιστεί εδώ ότι νέε χώρες μέλη πρέπει να προστίθενται εφόσον η... υπάρχει διαδικασία για αλλαγές μόνο όταν αυτό αφορά το πρώτο τμήμα. Και πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας ε, βέβαια τι συμβαίνει και στην περίπτωση που κάποιο άλλο κράτος θέλει να ενταχθεί στο δεύτερο τμήμα. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν κάποιες ασθένειε που επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο του ασθενεί, Για παράδειγμα, ανάλογα με το φύλλο του ή ανάλογα με την ηλικία του. Επιτάτες και γυναίκες αντιδρούν διαφορετικά στα φάρμακα. Για να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι είναι κατάλληλα τα φάρμακα για τους ασθενείς για τους οποίους προορίζονται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτές οι διαφορές να λαμβάνονται υπόψη στις κλινικές δοκιμές. Επίσης, αν υπάρχουν ε, κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και αυτά πρέπει να αναφέρονται πάντα για την ε, σύμφωνη γνώμη τώρα. Όσον αφορά το κεφάλαιο 5 του κανονισμού που αναφέρεται στη διαβούλευση, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τα μέλη που θέλουν να συμμετέχουν στις ε, κλινικές αυτές δοκιμές πρέπει να δίνουν ρητά τη σύμφωνη γνώμη τους. Θέλω να πω και δύο λόγια τώρα για την διαφάνεια. Σίγουρα πολλοί από τους συναδέλφους τα έχουν σκεφτεί αυτά. Εγώ δεν προτείνω σημαντικέ αλλαγέ στο κείμενο τη Επιτροπής. Αυτό όμως που λέω είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση για την πρόσβαση των χωρών στην, στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δοκιμές αυτές. Να λάβουμε υπόψη μας ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες οι οποίες επιτρέπουν το απόρριτο και πρέπει επίσης να βρούμε λύσεις για να βελτιώσουμε την διαφάνεια όσον αφορά τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Πολλοί παράγοντες που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό κόσμο ζητούν πλήρη πρόσβαση. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο στα αποτελέσματα, αλλά όχι κάτω από οποιαδήποτε προϋπόθεση. Να αποφύγουμε τα εμπορικά συμφέροντα. Γι' αυτό έχω επιφυλάξεις κατά πόσο και σε τι βαθμό πρέπει να είναι απόρριτα τα αποτελέσματα. Εξού και οι τροπολογίες που προτείνω και ό,τι άλλες τροπολογίες έχετε για το θέμα αυτό της διαφάνειας είναι ευπρόσδεκτες. Αυτό το οποίο, μάλλον υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν έχω αναφέρει, αλλά καλύτερα να μιλήσουν οι σκιώδεις συζητητές τώρα και μετά να συζητήσουμε εκτενέστερα ό,τι θέλετε σε κάποια επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας ή με τους ε, σκιώδεις εισηγητές εφόσον έχουμε τέτοιες συναντήσεις μαζί. Να πω τώρα για το χρονοδιάγραμμα πρόεδρε ή μετά. Το έχω μπροστά μου, αλλά ε, πείτε το για να μπορέσουν και άλλοι να παρέμβουν η κυρία Λεγκρίπ, να πούν την απόψή τους γι' αυτό. Προτείνω 31 Ιανουαρίου, εξέταση των τροπολογιών, αν συμφωνεί και η γραμματεία, στις 20-21 Φεβρουαρίου, να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ε, στις 20 Μαρτίου και να ψηφίσει στις 21 Μαρτίου η Επιτροπή μας, γιατί η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, προβλέπεται για τις 24-25 Απριλίου. Και ανάλογα βέβαια με το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, η Ολομέλεια θα αποφασίσει μετά. Προθεσμία λοιπόν, όπω είπα και πριν, είναι 31η Ιανουαρίου. Good. Well, thank you very much indeed for your very Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για την ε, ανασκόψή σα που ήταν πολύ επαγγελματική. Δίνω το λόγο στην κυρία ε, και μετά οποιαδήποτε άλλα μέλη θέλουν να σχολιάσουν και στη συνέχεια θα καλέσω την Κομισιόν να σχολιάσει. Κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρου του συναδέλφου μου, Φιλίπ Ζεβά, σκιώδου συζητητή για την ομάδα μας ε, του ΕΛΚΑ. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι ο Φιλιπ Ζιβά υποστηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεδομένου ότι υποστηρίζει την ιδέα για κανονισμό και όχι οδηγία άμεσης ε, και υποχρεωτικής εφαρμογής. Αυτός ο κανονισμός θα επιτρέψει την ομοιομόρφη εφαρμογή της νομοθεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνάδελφος μου κ. Ζουβά χαιρετίζει τις προσπάθειες εναρμόνισης, τυποποίησης και απλούστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που όπως φαίνεται έχουν λάβει μέτρα για να βγούμε από το διέξοδο της ε, κλινικής έρευνας στην Ευρώπη. Σας υπενθυμίζω ότι υποφέρει οι κλινικές δικοπές στην Ευρώπη από διοικητικό άκθος, δυσκολία εξουσιοδοτήσεων, έβρεση συμμετεχόντων, απώλεια ανταγωνιστικότητας και διάφορα άλλα προβλήματα. Στο σύνολο, ο συνάδελφός μου, κύριο Ζουβά, υποστηρίζει το σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητή μας του Κριστιαν Μπουζεύ υπό το πνεύμα που το παρουσίασε σήμερα. Μερικά λόγια, αν με επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τους ορισμούς. Τροποποίηση του ορισμού της κλινικής δοκιμής. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα μετάφρασης στη γαλλική έκδοση, δυστυχώς. γιατί μιλάμε για τον ορισμό της κλινικής δοκιμής, καλό θα ήταν να μην υπάρχει λάθος μεταφραστικό, αφού αποτελεί την αφετηρία ουσιαστικά του κανονισμού και όλης της διαδικασίας. Όσον αφορά τα άτομα με ελλειπείς ικανότητες, αυτά τα, Μιλάμε για νομικώς ανίκανα άτομα όπως ανήλικοι, η υποκειδαιμονία και μετά υπάρχουν τα άτομα τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα συνένεσης εκ των πραγμάτων λόγω αλλίωσης των γνωστικών τους ικανοτήτων. Αυτές οι δύο κατηγορίες ατόμων, ανίκανων ατόμων, διαχωρίζονται στη γαλλική νομοθεσία και αυτό δεν συμβαίνει στον κανονισμό αυτό. Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί όσον αφορά τις κατηγορίες κλινικών δοκιμών. Ο Φίλιπ Ζουβά υποστηρίζει τη στρατηγική της Κομισιόν για τη δημιουργία δύο κατηγοριών κλινικών δοκιμών και να διεξάγονται η επιτήρηση και η παρακολούθηση δεδομένου του κινδύνου. Θα ήθελε να υποβάλει μια τροπολογία για την κατάσταση της κατηγορίας κλινικών δοκιμών χαμηλής παρέμβασης με ε, κλινικές δοκιμές χαμηλού κινδύνου, ελάχιστου κινδύνου για δύο στόχους. Να ανταποκριθούμε στον κύριο στόχο του σχεδίου κανονισμού, το να βασίσουμε τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία στον προσθέμενο κίνδυνο της έρευνας, δηλαδή η προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο και δεύτερος στόχος φαίνεται Θεωρεί αναγκαίο ο Φιλιπ Ζιβάν να ευθυγραμμιστούν οι διατάξει του σχεδίου κανονισμού με την συνθήκη του Οβιέδο, η οποία έχει επικυρωθεί από τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό το κείμενο περιλαμβάνει και ορίζει τον όρο του ελάχιστου κινδύνου, τη ελάχιστη επικινδυνότητας. Όσον αφορά τα ευάλωτα άτομα, τα σχέδιο κορονισμού δεν προβλέπει κάτι για τι κλινικέ δοκιμέ, για ευάλωτα άτομα όπω οι γυναίκε, για παράδειγμα, ή άτομα που στερούνται ελευθερία. Ελευθεριών, ο Συνάδελφο Ζουβά θα ήθελε να υποβάλει μια τροπολογία όπου θα διευκρινίζει ότι τα κρατημέλη μπορούν να προβλέψουν διατάξει που θα προστατεύουν περισσότερο τα ευάλωτα άτομα. Τώρα, τις κλινικές δοκιμές, για τι κλινικέ δοκιμέ σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκη θα ήθελε ο κ. Ζουβά μία διάταξη όπου θα υπάρχει προκαταρκτική ε, συνένεση του ασθενού σε περίπτωση σοβαρού ε, επεισοδίου ή ατυχήματος ε, που απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση. Να περιλαμβάνεται λοιπόν αυτή η η ειδική διάταξη για την εκ των προτέρων συνένεση υπάρχει στις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια. Ο Φιλίπ θα ήθελε να υποβάλει μια τροπολογία για κατάργηση τη συνθήκη όπου αυτέ οι κλινικέ δοκιμέ έκτακτη ανάγκη μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο για τις περιπτώσει ελάχιστη επικίνδυνοτητα. Ουσιαστικά, εάν αυτό δεν αλλάξει για πολλά κράτη-μέλη, η διάταξη ω έχει στην παρούσα φάση μέσα στον κανονισμό θα μπορούσε να αποτελέσει οπισθοχώρηση ουσιαστικά διότι θα αποκλεί όλες τις δοκιμές για τα κοινοτόμα προϊόντα όσον αφορά τις ε, επιτροπές ηθικής. Μετά από τις πολλές επιφυλάξεις του και μετά από πολλούς προβληματισμούς υποστηρίζει πλέον ο συναδελφός μου τη Γενική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να ε, συνεργάζονται μέσω ενός ε, τεχνικού δελτίου, μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης και μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, αφήνοντας μεγάλο περιθώριο ελιγμών στα κράτη-μέλη για την οργάνωση σε εθνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν δυνάμει τη αρχή τη επικουρικότητα, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αξιολογούν τα τμήματα 1 και 2 του φακέλου εξουσιοδότηση και να αποφασίζουν κατά πόσο θα διατηρούν το διαχωρισμό το σημερινό ε, Επιτροπή Ηθική και Εθνική Επιτροπή. Υπενθυμίζω ο συναδελφό μου ότι η οδηγία του 2001 είχε επικριθεί ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό το ρόλο τη ε, Επιτροπή Ηθική και τη Εθνική Επιτροπή σε θέματα κλινικών δοκιμών και είχε επισημάνει τον ε, τεράστιο διοικητικό φόρτο που απορρέει από αυτό. Ο Φιλίπ ε, Ζουβά ε, θα ήθελα να τηρείται η αρχή της επικουρικότητας και της ασφάλειας των ασθενών φυσικά. Η ασφάλεια των ασθενών πρέπει να παραμένει προτεραιότητα για μας. Ο Φιλίπ Ζουβά υποστηρίζει την πρόταση του Κριστιαν Μπουζό για επανενσωμάτωση της ηθικής πτυχής και της Επιτροπής Ηθικής αυτών των ορισμών στο σχέδιο κανονισμού ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε παρανόηση. Όσον αφορά τις δυνατότητες έφεσης για την ε, αξιολόγηση του τμήματος 2 της έκκλησης για να υπάρχει δυνατότητα για τον διαφημιστή να κάνει ε, έκκληση για την ε, αξιολόγηση του τμήματος 2 θα ήθελε να πλησιωθεί αυτή η διαδικασία έκκλησης σε πολύ μικρές χρονικές προθεσμίες, ώστε να μην ε, βαραίνει η διαδικασία εξουσιοδότησης. Τώρα, όσον αφορά την κατάρτιση των αρμόδιων αξιολόγησης του αιτήματο και εκεί θα υποβάλει μια τροπολογία ο συνάδελφος Ζουβά για να διευκρινίζεται η ιδιότητα αυτών των μελών. Θα ήθελε τουλάχιστον τα μισά μέλη να είναι ιατροί πτυχίου χιατρή, σύμφωνα με τα εθνικά δίκαιο ε, επαγγελματικού ή ε, επίπεδου, επίπεδου εμπειρίας επαρκούς ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο αυτό. Τα μισά τουλάχιστον μέλη. Τώρα όσον αφορά το νέο αίτημα, μετά από απόσυρση αίτηση εξουσιοδότηση υποστηρίζει ο συναδελφό μου τη διατάξη του άρθρου 13 όπω έχει όπου υπάρχει δυνατότητα νέας αίτηση μετά από απόσυρση Ωστόσο, θα υποβάλει μια τροπολογία όπου θα υποχρεώνει τους προφητές να διευκρίνουν τους λόγους απόσυρσης της αίτησης εξουσιοδότησης και τις τροπολογίες που γίνονται κατά τη νέα αίτηση σε σχέση με την αρχική εκδόση του πρωτοκόλλου. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα διαφάνειας, Φτάνω στο τέλος κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζουμε την διάταξη της Κομισιόν για περισσότερη διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ωφέλεια προς τον ασθενή σε αυτή τη συζήτηση. Μας φαίνεται περιττό και επικίνδυνο να δημοσιεύονται όλα τα μη επεξεργασμένα δεδομένα τα οποία μπορεί να είναι και αρκετά ευαίσθητα διότι μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Είναι μια ευαίσθητη πτυχή. Ο Φίλιπ θα ήθελε να προχωρήσουμε προς μια ισορροπημένη προσέγγιση σεβόμενη την ε, αξιοπιστία και τον απόρριτο χαρακτήρα των δεδομένων και την ασφάλεια των ασθενών. Ε, η Κομισιόν προτείνει την ασφάλεια των δεδομένων. Ε, ο Φίλιπ Ζουβά θα ήθελε δημοσίευση λεπτομερών στοιχείων όσον αφορά αριθμού θανάτων, νοσηλείας κτλ. Το τελευταίο σημείο που μου ζήτησε ο Φίλιπ Ζουβά να σας ε, κοινοποιήσω, να κοινοποιήσω στους συζητητές τα προθεσμίες για τις εξουσιοδοτήσεις. Δεν θα ήθελε ο να τροποποιηθούν οι προθεσμίες θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των κλινικών δοκιμών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Good. Well, thank you very much indeed uh, for... Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Έχουμε σημαντική ιατρική ομάδα ε, εδώ που εργάζεται σε αυτό το φάκελο. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Άντες Ρίς, δεν ξέρω αν έγραψα το όνομά του σωστά, Διευθύντη Δημόσιας Υγείας στην Τιτζισάνκο, να απαντήσει στα σχόλια που ακούσαμε από τον εισηγητή και τους πιο εισηγητές. Καλώς ορίστε στην Επιτροπή μας και έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Δ. Μπούσεφ, για την πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση που έχετε συντάξει. Ελπίζω να συνεχίσουμε με αυτό το άριστο πνεύμα συνεργασία σε αυτή την Επιτροπή, διότι οι κλινικέ δοκιμέ είναι μόλι ένα κομμάτι τη μεγαλύτερη εικόνα τη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, τη οικονομία, τη επιστήμη, τη έρευνα και τη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εργασίας μας ε, και όπως είπατε έχει χάσει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια το 25% των κλινικών δοκιμών στην επικράτειά της. Ελπίζουμε επίσης ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτού του σημαντικού κανονισμού κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία και ότι θα καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι οι λύσεις μας πρώτα απ' όλα προστατεύουν τους ασθενείς αλλά επίσης επιτρέπουν και τις κλινικές δοκιμές ε, περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως είπε ο κύριος συζητητής, λάβαμε μεγάλη υποστήριξη από τους ενδιαφερόμενους, ε, ε, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τις επαγγελματικές ενώσεις, επαγγελματίες και τη βιομηχανία επίσης. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για δύο σημαντικά ζητήματα που ανέφερε ο κύριος Μπουσόη. Το πρώτο σχετίζεται με τη διαφάνεια αναφέρθηκε και στο σχόλιο που υπόθηκε εκ μέρους του κ. Ζουβά. Η διαφάνεια των κλινικών δοκιμών είναι εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι. του Έχει αποτελέσει το αντικείμενο δημοσίων διαβουλεύσεων, δημοσίων συζητήσεων. Είναι σημαντικό η πρότασή μας να είναι φιλόδοξη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η βάση δεδομένων και η πύλη που προετοιμάζουμε θα είναι δημοσίως προσπελάσιμα, αλλά ταυτόχρονα, όπως αναφέρθηκε στα σχολεία του κ. Ζουβά, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει προστασία των προσωπικών δεδομένων. καθώς και των εμπόρικα απόρριτων πληροφοριών. και θα πρέπει να φροντίσουμε και το ζήτημα της προσβασιμότητας σε όλα τα πρωτόκολλα. Εκεί τίθεται το ζήτημα του πόσες πληροφορίες μπορούμε να έχουμε δημόσιες προσπελάσιμε, α πούμε, για ανάλυση. Ε, θα θέλαμε επίσης να συζητηθεί το ζήτημα της ε, σύνοψης που θα δημοσιεύεται σύμφωνα με την πρόταση και όπως έχω ήδη αναφέρει είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Πόσα στοιχεία θα αποκαλύπτουμε σε αυτή τη σύνοψη για να βοηθούν την ανάλυση των ερευνητών και των ενδιαφερομένων. Προς ενημέρωση της Επιτροπής θέλω επίσης να πω ότι μόλις δημοσιεύσαμε στον ιστοτοπό μας ε, τις κατευθυντήριες γραμμές που αναπτύξαμε μαζί με τον Ευρωπαϊκό Ιατρικό Οργανισμό για τις πληροφορίες που θα παρέχουμε στον τρέχοντα κανονισμό μετά από την ολοκλήρωση των κλινικών δοκιμών σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ίδιο μοντέλο για τους μελλοντικού κανονισμούς. Ήθελα να τονίσω επίσης τέτοιου είδους κατευθύντηρες γραμμές έχουν αναπτυχθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου διότι Φυσικά μιλάμε για έναν τομέα παγκόσμιας εμβέλειας. Ε, ε, ε, το ίδιο συμβαίνει και στη ΣΥΠΑ, από τον FDA στις κλινικές, στο Μητρό Κλινικών Δοκιμών εκεί, του FDA. Άλλα σημαντικά ζητήματα είναι το ηθικό ζήτημα. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρόταση της ε, Επιτροπής ε, δεν αποσκοπεί να καταργήσει την Επιτροπή Ηθικής. Ο τρόπος που καταλαβαίνουμε ότι είναι περίπλοκη κατάσταση με όλα τα κράτη-μέλη και η αρχή της επικουρικότητας σε αυτόν τον τομέα και όπως ε, ανέφερε και ο κ. Μπουσόη, το σύστημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο σε ορισμένα κρατημέλη. Θέλουμε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν το ρόλο τους τα κρατημέλη σε αυτό το τομέα, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελα να δηλώσω ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο εξήγηση αυτής τη παρεμηνία, αυτή την πρόταση. Και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε προτάσεις που θα βοηθήσει την καλύτερη επεξήγηση, κατανόηση αυτής της ε, πρότασης, ώστε να αποφεύγονται οι παρανοήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, διότι νομίζω ότι η Αναμπίλεν θέλει να μιλήσει εκ μέρους του κ. Μακάρθη, που είναι σκιώδης. Ξέρω ότι έχετε κάποιες σημειώσεις μαζί σας, αν θέλετε λοιπόν να μας παρουσιάσετε κάποια σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω είπατε εκ μέλους του ECR τη κυρία Μακλάρκιν, σκιώδη του ECR που ζητά συγγνώμη που δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με την σημαντική εκθέση του κύριου Μπουσόη. Η ΕΜΑ χαιρετίζει την έκθεση τη Κομισιόν για την αναθεώρηση τη οδηγία για τι κλινικέ δοκιμέ, Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που έχουμε την ευκαιρία να υποβάλουμε μια γνωμοδότηση για αυτή την έκθεση της ΕΜΒΗ. Πρώτα απ' όλα, η ΕΜΑ θεωρείται από την τρέχουσα οδηγία. Μάθαμε ότι χρειαζόμαστε σαφήνεια των ορισμών. Πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και να μειώσουμε το κόστο και το φόρτο για τι βιομηχανίε. Χρειαζόμαστε ένα κανονισμό που θα ενισχύει ε, το ε, πόσο ελκυστικό θα είναι το περιβάλλον για την εξαγωγή κλινικών δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΕΜΑ λοιπόν θεωρεί ότι ο πρώτονόμονο κανονισμό θα μειώσει το διοικητικό αχθό για του ερευνητέ και του χορηγού μέσω της ε, εισαγωγής μιας προσέγγισης ε, ελάττωσης της επικινδυνότητας ώστε να δημιουργηθεί ένα καλύτερο περιβάλλον για την εξαγωγή των κλινικών δοκιμών. Έχει κάποια σχόλια για το σχέδιο γνωμοδότησης που θα ήθελα να αναφέρω. Είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη με την αναφορά στις ηθικές πτυχές της αξιολόγησης όπως αναφέρεται στην τροπολογία 11 του σχεδίου γνωμοδότησης. Ωστόσο, θεωρεί το άρθρο 7 δεν είναι το σωστό σημείο για κάτι τέτοιο, διότι αναφέρεται στην αξιολόγηση του τμήματο 2 μόνο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι Επιτροπές Ηθική αξιολογούν πτυχές και του τμήματο 1. Ω εκ τούτου, ε, θεωρεί ότι μια σαφή αναφορά θα ήταν προτιμότερη. Επιπλέον στην τροπολογία 14 του σχεδίου γνωμοδότηση, η ΕΜΑ πιστεύει ότι μέσω αυτού του τροποποιημένου ορισμού του ασθενούς θα είναι δύσκολο αν όχι αδύνατον να βρεθεί ένας κατάλληλο ασθενή ο οποίος θα είναι αντιπροσωπευτικό για μια ασθένεια μια οικογένεια ασθενειών στο διάστημα εφαρμογής του κανονισμού για σπάνιες ασθένειες αυτό μπορεί να φέρει σε διέξοδο την εξοδότηση, την άδεια κλινικών δοκιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το 19, στην τροπολογία 19, όπου έχουμε προσθέσει τη λέξη η αίμα δεν είναι σίγουρη αν οι δύο αυτές λέξει σημαίνουν το ίδιο. Κατά την άψη τη, το severity, που ήταν η προηγούμενη λέξη, αφορά κάτι μοιραίο που απειλεί τη ζωή. Αυτό θα ήταν μια ερώτηση που καλό θα ήταν να υποβάλουμε στην υπηρεσία γλωσσομαθονομικών ή ενδεχομένως η Κομισιόν θα μπορούσε να μας το διευκρινίσει. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσουμε την Κομισιόν για την πύλη που πρόκειται να εξυπηρετήσει για τις εφαρμογές. Λειτουργεί, είναι μια που μια εφαρμογή που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να δημιουργηθεί και πότε θα ανοίξει σε αυτή την περίπτωση. Πιστεύει ότι χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες για να δούμε την πρακτική πτυχή της πρότασης Τέλος, δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσο η εναρμόνιση των κανόνων για τη διεξαγωγή μη διασυνοριακών δοκιμών είναι αιτιολογημένη. Θα θέλαμε περισσότερες διευκρινήσεις για αυτό το σημείο. Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για να αναφέρουμε ότι μόνο οι εθνικές δοκιμές έχουν κινδύνους για τους συμμετεχόντες και ότι θα βελτιωθούν μετά από την ε, εφαρμογή των νέων αρμονισμένων κανόνων. Η ΕΜΑ επιθυμεί να συνεργαστεί με τον κύριο Σιγητή και τους Κιώδης για τη σύνταξη της παρουσίας νομοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much, uh, um, so, Christian... Ευχαριστούμε πολύ, Κρίστιαν ε, Ποζόη. Θα ήθελες να συνοψίσεις και ήθελες να Αναφέρεις άλλα ζητήματα. Έτσι μία κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες που περιγράφηκαν σήμερα και ευχαριστώ και για τα σχόλια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξαιρετική του συνεργασία θα ήθελα να του συγχαρώ ξανά για την εξαιρετική του πρόταση. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τόσο εξαίρετου ε, επαγγελματίες, με τόσο μεγάλη εμπειρία στον τομέα των κλινικών δοκιμών όπω τον κύριο Ζουβά. Είμαι μάλιστα περισσότερο από που υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι σκιώδης που έχουν πολλές καλέ ιδέε βελτίωση του κειμένου. Σήμερα έλαβα ε, είδα πολλές, άκουσα πολλές ενδείξεις για πιθανές τροπολογίες και κάποια σχόλια για τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Θα τα λάβω υπόψη και όταν συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες ε, θα κάνω και άλλα σχόλια πριν καταλήξουμε στις συμβαστικές για όλες αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ και πάλι. Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πολύ λοιπόν και για όσους συμμετείχαν. Προχωρώ τώρα στο τελευταίο θέμα της σημερινής διάθεσης. Α, παραπιπτόντως, ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήταν παρούσα εδώ. Λοιπόν, τελευταίο θέμα σημερινής σημερινής διάταξης. Ε, καλούμε εγώ ως εισηγητής να κάνω ε, την εισαγωγή για τον ε, τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων δεν ξέρω ποιος κοιόδης είναι εδώ. Ο κύριος Σμιτ, είστε εδώ ως Σάντου. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ο κύριο Σμιτ και εγώ θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι, πρόκειται σήμερα για την πρώτη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την πρόταση. Ήδη βεβαίω έχουν γίνει αρκετέ συναντήσεις. Θα δώσω το χρόνο στους εκπροσώπους Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ για θέματα υγείας να αποχωρήσουν. Λοιπόν, ο κύριος Σμιτ και εγώ θα κάνουμε την εισαγωγή, δεν ξέρω, ο κύριο Βαντερκάμπ είπε ε, ότι θα ήθελε να είναι παρόν, δεν είναι, λόγω καιρού ενδεχομένω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριο Σονίδη από την Κομισιόν, πολύ ωραία λοιπόν. το Συμβούλιο δεν ξέρω ποιον εκπροσωπείται για το θέμα αυτό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω πρώτα-πρώτα κάποια γενικά σχόλια. Να πω πρώτα-πρώτα ότι η έκθεσή μου ε, θα είναι, δεν θα είναι έτοιμη πριν από τις 20 Φεβρουαρίου. Σήμερα κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να μας κάνει η Κομισιόν μια παρουσία της αξιολόγηση επιπτώσεων. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται για όλα τα θέματα, αλλά εδώ χρειάζονται. Ε, εγώ είδα τη δική μας, αν θέλετε, αξιολόγηση επιπτώσεων και είδα και εσείς τι έχετε κάνει και το τον υπολογισμό κόστους κόστους-οφέλους. Θα θέλαμε λοιπόν να οργανώσουμε μια συνάντηση για να κουβεντιάσουμε ακριβώς τα θέματα αυτά. Ε, αιτιολογείτε επίσης την, ε, την πρότασή σας ε, για ομοιόμορφους τεχνικούς ελέγχους μάλλον εναρμόνιση αν θέλετε τεχνικών ελέγχων με στοιχεία κόστους κοίταξα τα στοιχεία ε, εγώ δεν είμαι σίγουρος όμως ότι συμφωνώ μαζί σας κι άλλο ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω Εγώ νομίζω όπως και για άλλες εκθέσεις και για άλλα θέματα ιδιαίτερα που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές και αυτό το θέμα ενδιαφέρει σαφώς τους καταναλωτές νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ζητούμε maximum εναρμόνιση αν υπάρχουν συστήματα τα οποία λειτουργούν ικανοποιητικά, που τελικά ε, ε, ε, εξυπηρετούν τους καταναλωτές και γίνονται αν θέλετε τεχνική έλεγχοι και ο τεχνικός έλεγχος τελικά είναι ένα θέμα για την ικανότητα των αυτοκινήτων να κυκλοφορούν σε ιστορικό επίπεδο δεν κυκλοφορούν τόσα πολλά στο εξωτερικό. Όταν λοιπόν έχουμε συστήματα τέτοια τα οποία λειτουργούν ικανοποιητικά, ε, κατά την άποψή μου ε, είναι ίσως υπερβολικό να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Δεν ξέρω δηλαδή σε τι θα ωφελούνταν ο καταναλωτής. ε, ε Έχουμε συστήματα όπου οι έλεγχοι γίνονται Ε, ε, ε, υπάρχουν χώρες τις οποίες ο τεχνικός έλεγχος γίνεται από μόνο αποκλειστικά από κρατικούς φορείς. Σε άλλες χώρες γίνεται από ανεξάρτητα από συγκεκριμένα συνεργεία αυτοκινήτων, ιδιωτικά εν πάση περιπτώσει. Ε, εδώ έχω την εντύπωση ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τα μοιραία ατυχήματα, ε, δηλαδή ουσιαστικά τη συμπεριφορά αυτών των οχημάτων στο δρόμο, είναι διαφορετική από ό,τι θα περμέναμε. και δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία που να κάνουν τέτοιου είδους συγκρίσεις δεν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι αν έχουμε ικανοποιητικά συστήματα θα πρέπει να τα αλλάξουμε τελείως και να τα ομογενοποιήσουμε τρόπον την Εκείνο που παίζει ρόλο είναι η συντήρηση των οχημάτων και όχι το ποιο κάνει τον τεχνικό έλεγχο. Θα έλεγα εγώ παραδείγματος χάρη. εγώ βέβαια έχω εμπειρία μοναχά από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά φαντάζομαι ότι ε, μπορεί να ισχύει και άμα γνώριζε κανείς όλα τα συστήματα που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Εγώ πάντως από την εμπειρία μου στον Ευρώπη Βασίλειο δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη η πλήρης εναρμόνιση εδώ. Βεβαίως θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο πάει πάρα πολύ αργά. η Κομισιόν ασχολείται βεβαίως και για τη μεταφορά η μεταβίβαση των οχημάτων από μία χώρα σε άλλη διαφορετική από αυτή στην οποία θα ξενομηθεί το όχημα. Λοιπόν, ε, εδώ ίσως καθυστερούμε εμείς. Το Συμβούλιο όμως ε, έχει εδώ προτείνει λύσεις πολύ πιο πολλέ πριν να αρχίσουμε εμείς ουσιαστικά τη δουλειά μας. Γιατί σε ορισμένα θέματα λοιπόν ε, έχει πολλέ αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις και ανησυχείς ε, το Συμβούλιο δηλαδή τα κράτη-μέλη ενώ για τούτο εδώ το θέμα που συζητούμε το τεχνικό άλλακο δεν ενδιαφέρεται ίσως ε, αυτό αντικατοπτρίζει κάπω την πραγματικότητα. Θα ήθελα όμω και τα στοιχεία τη Κομισιόν για να δούμε αν μπορούμε μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα αν έχετε συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά προς το παρόν εγώ λέω ότι δεν φαίνεται το θέμα αυτό να είναι επίγον για τους καταναλωτές. Τέλος πάντων, είμαστε επί αυτή όχι μόνο για την εσωτερική αγορά αλλά και την προστασία των καταναλωτών. Λοιπόν, δείτε, στο σκόρμπο του 2012 τα η αγορά των μεταχειρισμένων βρίσκεται στον Αδύρ για τρίτη, φαίνεται ότι βρίσκεται στον Αδύρ για τρίτη χρονιά ε, ξέρω ότι η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ασχολείται με το θέμα αυτό για να δει γιατί λόγω της συμπεριφορά των οχημάτων που θέτουμε στον δρόμο. Εκείνο όπως σας είπα που είναι ενδιαφέρον είναι η συντήρηση του αυτοκινήτου και με αυτή την έννοια ίσως και τα συνεργεία ε, τα οποία επισκευάζουν χειρισμένα αυτοκίνητα. Ε, η, παρακολούθηση αν θέλετε των, ε, των χιλιόμετρων ή των μιλίων που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο ή καταγραφή των, των μιλίων που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο. Ε, έχω την αίσθηση δηλαδή ο ότι ο ετήσιος τεχνικός έλεγχος ε, δεν ε, ε, έχει τόσο μεγάλη επίπτωση στο ούτε, κα, ούτε συμπεριφορά του οχήματος και άρα στο αριθμό των ατυχημάτων ούτε στο πώς ε, ούτε στην αγορά μεταχειρισμένων ή όχι αυτοκινήτων είναι μικρή η επίδραση του τεχνικού ελέγχου εκείνο που ενδιαφέρει είναι η συνεχής παρακολούθηση και συντήρηση Τώρα βέβαια βλέπουμε να έρχονται από τη Γαλλία πελάτες να αγοράζουν τα χειρισμένα αυτοκίνητα στο Βέλγιο. γιατί, επειδή η αγορά είναι πιο αξιόπιστη στο Βέλγιο. Μπορεί. Θέλω να πω, τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι η Κομισιόν έχει απόλυτο δίκιο στην αιτιολογία της, για την ε, υποβολή της πρότασης αυτής. Εγώ σε γενικές γραμμές συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι δεν μας χρειάζεται κανονισμός προφανώς, διότι δεν είμαστε υπέρ της maximum εναρμόνισης. Εγώ θα έλεγα ότι πράγματι καλύτερα είναι να προβλέψουμε οδηγία εδώ, αν θέλουμε οπωσδήποτε νομοθετική πράξη. Το πιο σημαντικό όμως για μας είναι η αναγνώριση τύπου και οι τεχνικές πληροφορίες. οι τεχνικές πληροφορίες είναι απαραίτητες, δεν το συζητώ. Όμως θέλουμε επίσης την πρόταση αυτή να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες αυτές θα δίνονται και στα συνεργεία εκείνα τα οποία ε, συντηρούν ή επισκευάζουν τα οχήματα. Θα πρέπει να δίνει ο κατασκευαστής τα στοιχεία αυτά. πληροφορίες ίσως και παραπάνω από αυτές που σχετίζονται με τα καυσαέρια. Τον έλεγχο των καυσαρίων. Εσείς προτείνετε να έχουμε μία πύλη δεδομένων για τα στοιχεία ε, για τους ε, αυτούς που κάνουν τους ελέγχους ή ε, θέλουμε για τα καινούργια συστήματα και τα λοιπά, για τα βέλτιστα συστήματα. Με αυτή την έννοια προωθείται και επενδύσει για τα καινούργια συστήματα. Αυτό δεν ξέρω με βρίσκει σύμφωνο. Και μιλάτε και για τους ελέγχους στο μέλλον. Δείτε, ούτως ή άλλως, τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται τώρα ε, ή που θα κατασκευάζονται στο μέλλον θα έχουν ενσωματωμένα συστήματα διαγνωστικά. Ε, ε οπότε δεν ξέρω, ε, τι να σας πω, δεν ξέρω αν χρειάζεται να αλλάξουμε το σύστημα. Θα υπάρχουν διαγνωστικά συστήματα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. και άπαξ και εγκριθεί το συγκεκριμένο όχημα, ο συγκεκριμένο τύπο, τότε και τα αποτελέσματα του διαχρονογνωστικού συστήματο θα είναι έγκυρα. Άμα λοιπόν έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο δουλεύει σωστά, και κάνει σωστά τη διάγνωση ας το πούμε για οποιαδήποτε ε, προβλήματα ή για τη σουσπανσιό είτε για, το, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου και τα λοιπά, τότε ε, αυτά ενδεχομένω μας καλύπτουν και θα πρέπει να γίνει και μια αναθεώρηση στο μέλλον αυτών των τεχνικών ελέγχων. Είναι σημαντικά όλα αυτά, δεν το αμφισβητώ. Θα πρέπει να δούμε και για την ανάρτηση που ανέφερα πριν, ε, τα καινούργια συστήματα ηλεκτρονικά Και, τα λοιπά, και πώς σχετίζονται με την πρόταση που κάνετε. Αλλά ουσιαστικά αλλά επίσης, θα πρέπει να δούμε και τη σχέση μεταξύ αναγνώριση τύπου και των επιδόσεων. υποβάλλεται το συγκεκριμένο όχημα για έλεγχο και βγαίνουν ορισμένα αποτελέσματα. Το κατά πόσον αυτά τα αποτελέσματα είναι ακριβώς αυτά τα οποία υπήρχαν και βάσει των οποίων έγινε η αναγνώριση τύπου δεν ξέρω αν είναι και το, μα, το απόλυτο που πρέπει να ζητήσουμε ή αν αυτό ουσιαστικά προσδιορίζει το κατά πόσον είναι κατάλληλο για να κυκλοφορήσει στον δρόμο το όχημα. Μπορεί κανείς να έχει αλλάξει, ξέρω, τον κινητήρα και αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και το θέμα για τα λεγόμενα ιστορικά οχήματα τώρα και από αυτό το συγκεκριμένο το θέμα αυτών των αυτοκινήτων θα πρέπει να ανατεθεί πλήρως στα κράτη-μέλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πράγματι απαλλάσσει από το τεχνικό έλεγχο τα οχήματα που είναι άνω των 30 ετών. Με, γιατί, διότι προποθέτει ότι θα είναι αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία είναι αντίκα θα τα παρακολουθεί κάποιος άλλος θα τα φροντίζει κάποιος συλλέκτης. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν να το δούμε. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτηματικά που έχω. Θα δούμε μαζί με τον εισηγητή τι θα κάνουμε. Ε, θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο παραπάνω για την αγορά των μεταχειρισμένων οχημάτων γιατί σας λέω ότι και άλλες γενικές διευθύνσεις όπως η ΣΑΝΚΟ ασχολείται με αυτό βεβαίως όχι μόνο από την οπτική γωνία των τεχνικών ελέγχων αλλά από και από άλλες κοπιές ε, αυτά από πλευράς μου ε, να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σμιτ και μετά να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα σας μιλήσω και για τις προθεσμίες που κατά Σμιτ αντί καθιστώ τον κύριο Μάντερς, ο οποίος πρέπει να πάει στον... Ε, ο οποίος θα πάει στο νοσοκομείο. Θα ήθελα να πω απλά... More comments from, from Tuan and then I... Θα ήθελα να πω απλά ότι υπάρχουν πολλά <laughs> ε, ερωτηματικά εδώ. Παρεμπιπτόντως εγώ έχω κταίω τεχνικό έλεγχο αύριο, ε. Αλήθεια. Η Κομισιόν έχει υποβάλει μια καλή πρόταση και γι' αυτό ο κ. Μάντερ συμφωνεί με τα περισσότερα από αυτά που προτείνονται. Είναι κατά της πλήρους ε, εναρμόνισης των τεχνικών ελέγχων, είναι υπέρ της αμοιβαίας αναγνώρισης όμως των ελέγχων αυτών. Φαντάζομαι ότι πολλές από τις παρατηρήσεις που έκανε ο πρόεδρος θα μπορούσαν να βρουν σύμφωνο και τον κύριο Μάντερς. Εν πάση περιπτώσει, στη χώρα μου να σας πω εγώ προσωπικά τώρα, ξεκινήσαμε τους ελέγχους αυτούς το 1963 και μετά ιδιωτικοποίησαμε το όλο σύστημα, δηλαδή δώσαμε τη δυνατότητα σε ιδιωτικά συνεργεία να κάνουν τους ελέγχους αυτούς. Παλιότερα όταν κάθε φορά που έπρεπε να περάσω κταίο, επειδή είχα δεύτερο χέρι αυτοκίνητο ή δεν είχα λεφτά να πάρω καινούρια, ή ένιωθα σαν να πήγαινα στον οδοντίατρο. Δεν χρειάζεται φαντάζομαι να πω πολλά πράγματα, δεν καταλαβαίνετε πως αισθανόμουν. Δεν ξέρω, ίσως ισχύει το ίδιο και τώρα, αλλά τότε, τότε πραγματικά είχα την αίσθηση ότι πήγαινα σε μία αρχή η οποία θα έκανε τον έλεγχο, τουλάχιστον στη χώρα μου. Δεν ξέρω, τώρα ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα, ίσως στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην υπάρχει η αίσθηση της εξουσίας της αρχής αν θέλετε. Μάλκολμ Χάρμπορ μίλησες για κανονισμό ή οδηγία. Το κουβέντιασα αυτό και με τον κύριο Μάντερς, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα τους κανονισμούς. Εγώ αντιθέτως δεν τους αγαπώ. Και η ιστορία μας δείχνει ότι ιδιαίτερα την σήμερον ημέρα η εναρμόνιση στην Ευρώπη όταν έχουμε 27 κράτη-μέλη είναι λίγο δύσκολη. Θα πρέπει να δίνουμε κάποιο περιθώριο ευελιξία για τα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν λέω σε κάποια μέρη της Ευρώπης απαιτείται κανονισμός. Γιατί είναι τα κράτη-μέλη κακά και δεν εφαρμόζουν καλά τις οδηγίες. Εγώ όμως προέρχομαι από μια χώρα η είναι αρκετά αυστηρή στην εφαρμογή των κανονισμών, των οδηγιών κτλ. Ε, Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε το θέμα και από τη σκοπιά του καταναλωτή. Ε, για τον καταναλωτή είναι λίγο... δεν είναι και πολύ σεξι η πρόταση αυτή. Είναι μάλλον βαρετή. Ε, υπάρχει όμως ενδιαφέρον και παρεμπιπτόντως να πω ότι είμαστε πολύ λίγοι εδώ στην αίθουσα. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί αρχίσαν να διοικούν τον κόσμο και έχουν δουλειές αλλού και όχι στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, τι ενδιαφέρον επιδεικνύεται από τη μικρή παρουσία μελών εδώ στην Επιτροπή δεν ξέρω. εγώ συμφωνώ ότι χρειάζονται ελάχιστα πρότυπα. Αυτό είναι σίγουρο. Minimum standard, ναι. Στη χώρα μου το συζητήσαμε το το θέμα αυτό, ιδιαίτερα σε σχέση με τα φορτηγά, τα οποία σε αντίθεση με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν έρθετε στο Τρέλεμποργκ το ferry boat με τα φορτηγά και εγώ πάω στο εξοχικό μου βλέπω τα φορτηγά αυτά τα τεράστια τα γιγαντιαία και λέω Παναγία μου τουλάχιστον έχουν καλά φρένα λειτουργούν σωστά να είναι ασφαλή βεβαίως αυτό είναι θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το συζητώ αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα. για τα ιστορικά οχήματα. Γιατί και στο δικό μου το γραφείο ε, κάποιοι έθεσαν τα ερωτήματα. 30 χρόνια μας είπατε εσείς, ηλικία 30 ετών. Εσείς τώρα το αλλάζετε αυτό και αναφέρεστε στη μερομηνία κατασκευής. Ήρθαν σε επαφή μαζί μου κάμπος οι καταναλωτές όπως σας είπα και μου είπαν ότι η ιδέα εδώ ότι ουσιαστικά οι αντίκες ή τα ιστορικά οχήματα δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις αυτές. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λοιπόν. Ε, σας διαβεβαιώ πάντως ότι διαβιβάσω όλα τα σχόλια που γίνονται εδώ στον Μάντερς. Ναι, θα συνεχίσουμε να δικούμε τον κόσμο εμεί πάντω, λέει ο κ. Χάρμπορ. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα και μετά θα συνεχίσουμε με τα διάφορα σημεία. Παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι ενδιαφέρεται όλο ιδιαίτερω για την πρόταση αυτή και μάλιστα όλο και περισσότερο μια που έχουμε την τύχη να έχουμε ως εισηγητή κάποιον που είναι ειδικό στα οχήματα. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε να έχουμε την ίδια επικοδομητική σχέση όπως είχαμε και μέχρι τώρα για το e Η πρόταση αυτή είναι λοιπόν μια σημαντική πρόταση στα πλαίσια γενικότερα της πολιτικής μας για την οδική ασφάλεια είναι πράγματι πολύ σημαντικό και μαθαίνουμε πολλά δουλεύοντας μαζί σας για μια τέτοια πρόταση προκειμένου να ε, συμπεριλάβουμε περισσότερο τον παράγοντα καταναλωτής. Νομίζω ότι θα δεχτώ την πρόσκληση του Προέδρου, εφόσον έχετε χρόνο δηλαδή, να σχολιάσω για την ε, μελέτη επιπτώσεων. Είτε εδώ, είτε στην... πριν πάτε στην Ολομέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια η ασφάλεια και πρέπει να ξέρετε ότι παρόλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, είναι δύσκολο να εκφραστεί ποσοτικά. Προσπαθούμε λοιπόν να βασιστούμε σε αντικειμενικά δεδομένα και όσο γίνεται περισσότερο σε ό,τι γνώση διαθέτουμε τη συγκεκριμένη στιγμή του χρόνου. Πρόλευση της πρότασης αυτής είναι ότι εξακολουθούμε να δουλεύουμε βάσει της οδηγίας, η οποία τώρα από τεχνική άποψη έχει φτάσει τα δέκα έτη ζωής. Και το γνωρίζει πολύ καλά και ο πρόεδρος ότι τα οχήματα έχουν τροποποιηθεί πολύ, έχουν αλλάξει πολύ και μαθαίνουμε από τις αλλαγές οι οποίες έχουν εισαχθεί στις χώρες μέλη. Συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας όλο και περισσότερο που έχουμε να υπάρχουν από τρίτα μέρη δοκιμές για συγκεκριμένα είδη οχημάτων. Επ' αυτού λοιπόν πρέπει να είσαστε σίγουροι για το ότι η πρότασή σας δεν αποτελεί φραγμό στην επιλογή των κρατών μελών να ενισχύσουν το ένα ή το άλλο είδος δοκιμής ή οργανισμού που κάνει τις δοκιμές. Βέβαια, πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από ποτέ στην ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρεται. Και ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να ανανεώνουμε κάθε τόσο τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέλουμε. Συνεπώς, Εάν έχετε την εντύπωση ότι αυτού του είδους η νομοθεσία, αυτή η πρόταση δηλαδή, θέλει να βάλει ανώτατες προδιαγραφές εναρμόνισης, να ξέρετε πως δεν είναι αλήθεια αυτό. Καθόλου. Συνεχίζουμε με την ίδια αρχή, η οποία είναι να βάλουμε τις προδιαγραφές που είναι αναγκαίες έτσι ώστε τα οχήματα να περνάνε από τη μία χώρα στην άλλη και νομίζω το παράδειγμα που δώσατε πριν από πέντε λεπτά είναι πάρα πολύ καλό. Συγχρόνως τα μεταχειρισμένα οχήματα αγοράζονται σε διαφορετικές χώρες μέλη. Γι' αυτό και λέμε ότι υπάρχει ευθύνη από όλες τις πλευρές και γι' αυτό ο, η πτυχή εσωτερική αγορά έχει πολύ μεγάλη σημασία στην πρόταση αυτή. Αυτό που περιμένουμε από εσά είναι να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε ενδεχομένω την πρότασή μας όσον αφορά το φιλτράρισμα. Τελικά ποιες θα είναι οι καλύτερες ελάχιστες προδιαγραφές από την εμπειρία που υπάρχει στα κράτη-μέλη, αλλά και βάσει βέβαια και της μελέτης αντικτύπου. Υπάρχουν και διάφορα πολύ σημαντικά στοιχεία στην πρόταση αυτή που έχουν ε, άμεση σχέση με τη δικιά σας τη δουλειά. Το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης, για παράδειγμα. Εμείς προσπαθήσαμε, αν μη τι άλλο, να συμπεριλάβουμε την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αλλά θα μπορούσε κανείς να πάει ακόμα πιο μακριά. Και αυτό είναι που περιμένουμε από εσά. Επίσης, στην πρόταση αυτή υπάρχει μια σχέση με... Και προσέξτε, αυτή την πρόταση εσείς δεν πρέπει να τη δείτε σαν μια υποχρέωση για να έχετε μια πλήρη απόδειξη για κάθε τροποποίηση που θα γίνεται στο όχημα. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας όμως είναι να δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται και να ζητήσουμε από τους επιθεωρητές να ελέγχουν κατά πόσο τα βασικά στοιχεία του οχήματος, για παράδειγμα το σύστημα τροχοπέδησης, έτσι, τα φρένα, χρειάζονται κάποια βελτίωση ή όχι. Επίσης, υπάρχει και συνδευτική πρόταση για βελτίωση της πληροφορίας των πληροφοριών που δίνουν οι αυτοκινητοβιομηχανείς σε αυτούς που κάνουν τους ελέγχους. Μια πολύ σημαντική πτυχή επίσης είναι η καταπολέμηση της απάτης. Αναφερθήκατε και εσείς σε αυτό, Πρόεδρε, και πολύ χαίρομαι που το είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για τον καταναλωτή. για τα παλιά ιστορικής αξίας ε, οχήματα, συλλογικής αξίας. Νομίζω ότι, συλλεκτική συγγνώμη νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε να μην δώσουμε τη στραβή εντύπωση, γιατί αυτό το οποίο εμείς στοχεύουμε είναι να προσφέρουμε περισσότερη ελαστικότητα από ό,τι το τρέχον σύστημα, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα των 30 ετών, να την έχουν τα κράτη-μέλη, αλλά και να εισάγουμε και μια ελάχιστη ρήτρα ασφάλειας, δηλαδή να λέει ότι τα ανταλλακτικά ή που πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή να είναι πολύ κοντά σε αυτά. Αυτή η δυνατότητα πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα αυτά δεν αποτελούν κίνδυνο στους δρόμους μας. Η φύση τώρα των ε, κέντρων ελέγχου. Είμαστε ουδέτεροι γι' αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό, το είπατε και εσείς πρόεδρε, αναφερθήκατε στα αποτελέσματα του βαθμολογίου. Είναι μια πρόσκληση προς εμάς να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το συνολικό και γενικό σύστημα επιθεωρήσεων τη στιγμή που τελικά η καλύτερη και μοναδική εγγύηση που έχει κανείς όταν αγοράζει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι το πιστοποιητικό. Η αξιολόγηση δηλαδή που κάνει στο όχημα το κέντρο αυτό. Γι' αυτό θα έλεγα ας δούμε τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα που έχει οδηγήσει στην πρόταση αυτή και από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί, να το ξέρετε, για κάθε συνεργασία μαζί σας ώστε να βελτιώσουμε παρετέρω την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για την επικοδομητική σας απάντηση. Θα προσπαθήσουμε να δούμε μήπως γίνει παρουσίαση αυτή είτε στους σκιώδες είτε σε ολόκληρη την Επιτροπή μας. Θα δούμε. Ευχαριστούμε που μας ε, επιβεβαιώσατε κάποιες από τις πτυχές που θέλαμε κι εμείς. Θέλουμε η συνεισφορά μας να είναι μια προστιθέμενη αξία. Και σίγουρα δεν θέλω να έχουμε επικαλύψεις με την επί της ουσίας αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην ακρόαση αυτή τη βδομάδα. Πρέπει να κοιτάξω το μαγνητοσκοπημένο βίντεο. Όπως βλέπετε πάντως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κύριο Σμιτ και εμένα κλπ. Λοιπόν, ε, σκοπεύω μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου να έχω ετοιμάσει το κείμενο και να το εξετάσουμε στις 20 Μαρτίου με προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 25 Μαρτίου. Να ψηφίσουμε εδώ στις 25 Απριλίου και έτσι προλαβαίνουμε και την ψηφοφορία που θα γίνει στην Επιτροπή Μεταφορών το Μάιο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και σας και τους συνεργάτες σας που ήρθατε από την γενική σας διεύθυνση. Είναι πολύ καλό που σας βλέπουμε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σμιτ που ήταν εδώ. Και έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας για σήμερα. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο πρόεδρος. Θα συνεδριάσουμε και πάλι το Φεβρουάριο. Από τις 20, ε, 20 δηλαδή και 21 του μηνός. Πρωί και απόγευμα και τις δύο μέρες. Και θα δούμε μήπως μπορούμε και να συνονεθούμε με την Επιτροπή Μεταφορών να κάνουμε κάτι μαζί. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όσους μας παρακολούθησαν στο διαδίκτυο. Έληξε η συνεδρίαση.